Okay, colleagues, um, we're going to make a start. Ξεκινάμε. Σημείο 1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνεται. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποια πρόοδο στο θεματολόγιο για τη μετανάστευση σήμερα το απόγευμα. Σημείο 2. Ανακοινώσει του Προέδρου. Ε, σε ό,τι αφορά το γλωσσικό καθεστώς ε, διερμηνία στα δανέζικα, λετονικά, κροατικά και ε, ιρλανδέζικα δεν είναι διαθέσιμη σήμερα το απόγευμα. Και μια άλλη ακόμα ανακοίνωση. Ο κύριος Κύρκος ε, πριν από τη συνεδρίαση ήρθε σε επαφή μαζί μου για να μου πει ότι υπάρχουν προβλήματα, ακόμα περισσότερα προβλήματα με τη μετανάστευση και το σύστημα μετανάστευση στην Ελλάδα, σημαντικά οικονομικά προβλήματα ε, που επηρεάζουν ε, τις, ε, την μετανάστευση στην Ελλάδα και είπε ότι θα μου στείλει και ένα email θα ε, η Γενική Διεύθυνση Home ε, Ιστορικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καλό είναι να δει αυτά τα θέματα. Ε, ακούω αρκετό θόρυβο, είσαστε λίγο άτακτοι σήμερα. είναι σημαντικό το θέμα αυτό, παρακαλώ πολύ. θα το συζητήσουμε και κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης και στους συντονιστές θα το θίξω εγώ αύριο. Το βασικό θέμα της Μέσης διάταξης σήμερα είναι το σημείο 3, το Ευρωπαϊκό Θεμετολόγιο για τη Μετανάστευση. Παρουσίαση ε, από τον Ματίας Ρούιτε, Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διευθύνσης Home της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με, τα, με τις προτάσεις, την πρόταση απόφαση Συμβουλίου σχετικά με τα προσωρινά μέτρα στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ελλάδας και της Ιταλίας. Ε, υπάρχει η, θα συζητήσουμε την, ε, το σχέδιο έκθεσης συγγνώμη, ε, επανέρχομαι στη σημείο 3 παρουσίαση καταρχήν του Ματία Ρούιτε για το θέμα της απόφασης συμβουλίου και μετά θα προχωρήσουμε στα υπόλοιπα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Είναι μεγάλη μου χαρά να σας ε, κάνω ένα, μια γρήγορη παρουσίαση του πακέτου, εφαρμοστικού πακέτου που υπέβαλε η Κομισιόν στις 27 Μαΐου του τρέχοντος έτους. Ο Επίτροπος ο κ. Αβραμόπουλος ε, σας παρουσίασε το συνολικό θεματολόγιο για τη μετανάστευση. Γνωρίζετε επίσης ότι προβλέπονται 50, πάνω από 50 δράσεις ε, ε, μέσα σε αυτό το πακέτο, σε αυτό το θεματολόγιο. Το πρώτο εφαρμοστικό πακέτο δημοσιεύθηκε μόλις 15 μέρες μετά τη δημοσίευση του θεματολογίου και ε, αφορά έξι κυρίως σημεία. Ένα από αυτά θα το συζητήσουμε αργότερα σήμερα. Να σας ε, πω δύο λόγια για το πρώτο θέμα στο οποίο πιο πολύ εστιάστηκαν τα μέσα ενημέρωσης που είναι ε, το θέμα της ε, ε, επανεγκα... μετεγκατάστασης, επίγουσας μετεγκατάστασης που είναι το τρίτο σημείο του πακέτου. Η δημόσια συζήτηση για την μεταναστευτική πολιτική επικεντρώθηκε πολύ σε νούμερα και ποσοστώσεις. Ενώ στην πραγματικότητα το θεματολόγιο για τη μετανάστευση είναι κάτι πολύ πιο πλατή, πολύ πιο ολιστικό, προσπαθεί να έχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες, ε, αφορά και την νόμιμη μετανάστευση. Πολλά από αυτά πνίγηκαν από την πολιτική συζήτηση των τελευταίων εβδομάδων εξαιτίας του ότι η κοινή γνώμη και η γενικότερο διάλογο συζητήθηκε στη, μετα... στη Ε, η δημοτική βάση είναι το άρθρο 78.3 της συνθήκης και προσπαθούμε μέσω αυτής πρότασής, να πρότασής μας να δείξουμε αλληλεγγύη προς την Ελλάδα και την Ιταλία μέσω ενός συστήματος επίγουσας επανεγκατάστασης 40.000 ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Ε, είπατε, μιλήσατε για την, ε, για την ο κ. Ε, το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι ότι ε, παρουσιάζεται μια σημαντικότατη αύξηση των ε, ροών αυθεντικών ετούντων άσυλο που φτάνουν μέσω της θάλασσας από την Τουρκία στα ελληνικά νησιά. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τρομακτικά προβλήματα ε, στην υποδοχή αυτών των ατόμων. Πάνω από 50.000 άτομα έφτασαν με αυτόν τον τρόπο τους τελευταίους μήνες στα νησιά του Αιγαίου. Και θα πρέπει να κάνουμε την διάκριση ανάμεσα στην, στην οδό έλευσης της Ανατολικής Ευρώπης και αυτήν της Τη Ανατολική Μεσογείου και αυτήν της Κεντρικής Μεσογείου στην οποία είχαμε εστιάσει την προσοχή μας στο παρελθόν. Οπότε προτείνουμε ε, να ε, επανεγκατασταθούν 40.000 άτομα που ε, χρήζουν διεθνούς προστασίας 24.000 από την Ιταλία και 16.000 από την Ελλάδα. Θέλουμε να δείξουμε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και ταυτόχρονα θέλουμε να ε, ε, πείσουμε τα κράτη-μέλη να αναλάβουν τις ευθύνες τους ό,τι αφορά ε, τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει για τη βελτίωση των συστημάτων μετανάστευσης και ασύλου. Ελπίζουμε ότι ε, το σύστημα αυτό θα υποστηριχθεί με 240 εκατομμύρια, 6.000 δηλαδή ευρώ κατάτομο που θα επανεγκατασταθεί. Και θα δημιουργήσουμε ένα σύστημα επιμελητίας ε, από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξη για το Άσυλο και άλλες ευρωπαϊκές υπηρεσίες. Η συζήτηση όπως σας είπα ήταν αρκετά ε, δεικτική ε, αλλά ε, το Συμβούλιο καθόρισε ένα συγκεκριμένο νούμερο. 40.000. Ε, διαφώνησε με την ε, Κομισιόν σε ό,τι αφορά το μηχανισμό, το Συμβούλιο, αλλά ε, ενέκρινε το νούμερο. Οπότε ε, αυτό αποτελεί δέσμευση και αναμένουμε εμείς ως Κομισιόν η δέσμευση αυτή να τηρηθεί. Ήδη σήμερα το πρωί μου σε επαφή με διάφορα κράτη-μέλη και συζητείται προφανώς η κλίδα ανακατανομής και περιμένουμε να δούμε αν τα κρατη θα τηρήσουν αυτή τη δέσμευση. Και εσείς φαντάζομαι θα συζητήσετε αυτό το θέμα με τους υπουργούς στο άτυπο συμβούλιο σε μερικές μέρες. Ως υποσημείωση υποσχεθήκαμε ότι θα υποβάλουμε ένα πιο μόνιμο μηχανισμό ε, επίγουσας μετεγκατάστασης μέχρι το τέλος του χρόνου. Και όταν υποβάλουμε αυτή μας την πρόταση θα συζητήσουμε όλα τα στοιχεία εν ευθέτω χρόνο. Τώρα, τι κάνουμε με τους 40.000. Ε, είναι ε, σαν ένας βραστήρας. Η, εμείς αυτό που δημιουργούμε είναι βαλβίδα διαφυγής. Ε, το μόνιμο σύστημα επανεγκατάστασης θα είναι μια βαλβίδα την οποία θα χρησιμοποιούμε κατά το δοκούν και δεν θα είναι απλώς μια επίγουσα βαλβίδα διαφυγής. και το τρίτο στοιχείο το οποίο θα συμπληρώσει το πανόραμα είναι ότι θα δούμε το συνολικό σύστημα για να δούμε αν δουλεύει. Αυτή τη στιγμή, ε, το, ενώ το σύστημα του Δουβλίνου, αλλά αυτή τη στιγμή με ελάχιστες εξαιρέσεις βρισκόμαστε εντός του συστήματος του Δουβλίνου. Τώρα, έχουμε υποβάλει ένα προτάσεις για ένα ευρωπαϊκό σύστημα επανεγκατάστασης ε, με 20.000 θέσεις για δύο χρόνια. Ελπίζουμε ότι τα κράτη-μέλη θα αναλάβουν συγκεκριμένε αριθμητικέ δεσμεύσεις για την εφαρμογή του. Ε, με την υπατή αρμοστία του για τους πρόσφυγες ε, θα χρηματοδοτήσουμε 10.000 με 10.000 ευρώ το κάθε άτομο που θα επανεγκαθίσταται. Και σε γενικές γραμμές αυτό το σύστημα είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος του σχεδίου δράση μας κατά της λαθρομετανάστευσης. Αν καταφέρουμε να διακόψουμε, μάλλον για να καταφέρουμε, να διακόψουμε ε, τους, μάλλον αν καταφέρουμε να διακόψουμε τους, τις οδούς ε, της λαθρομετανάστευσης θα πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους για να ε, δεχόμαστε ε, άτομα, μετανάστες. Ε, ο, ο ΙΕ πρότεινε 20.000 άτομα. Κάτι το οποίο θα εντάσσεται και στην Ατζέντα 2020. Σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της ε, λαθρομετανάστευσης ε, ε, των διακινητών, έχουμε διάφορες δράσεις σε τέσσερα κεφάλαια. Πιο ισχυρή αντίδραση πλευράς αστυνομίας και δικαστικών και δικαστικού συστήματος. Δεύτερον, βελτίωση της συλλογή και ανταλλαγής πληροφοριών σε στενή συνεργασία με την ε, αποστολή της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βελτίωση της πρόληψης ε, της λαθρομετανάστευσης και βοήθεια στους ευάλωτους μετανάστες και πιο ισχυρή συνεργασία με τρίτες χώρες. Αυτά είναι τα τέσσερα κεφάλαια. Να σας δώσω τώρα και ορισμένα παραδείγματα. Καταρχήν, θα δούμε ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διάφορες κυρώσεις που υφίστανται ε, να αποφύγουμε ε, την ε, καταδίκη, την, ε, κυρώσεις άτομα τα οποία απλώς βοηθούν ανθρωπιστικά τους μετανάστες. Δεύτερον, οι οικονομικές έρευνες προκειμένου να εντοπίσουμε και να κατάσχουμε ε, πόρους και χρήματα ε, των δικτύων διακινητών. Τρίτον, θα αναπτύξουμε τρόπους και ε, μέσα επικοινωνίας και θα προσπαθήσουμε να καταπολεμήσουμε τη λαθρομετανάστευση μέσω εξτρατιών ευαισθητοποίησης αλλά και αλληλοπληροφόρηση εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέταρτο στοιχείο, σε αυτό το πρώτο ε, εφαρμοστικό πακέτο και ήδη σας λέω ότι ετοιμάζουμε τα επόμενα εφαρμοστικά πακέτα. Ε, αυτό το τέταρτο στοιχείο είναι οι, οι κατευθύνες γραμμές της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε μια κοινή ευρωπαϊκή πρακτική για αυτό το θέμα. Ήδη έγινε στις 16 Ιουνίου μια πολύ χρήσιμη συνεδρίαση με τα κράτη-μέλη και νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε πως το έγγραφο αυτό που υποβάλαμε περιλαμβάνει τις καλύτερες, τις βέλτιστες ε, πρακτικές που θα πρέπει να εφαρμόζονται ε, σύμφωνα με τον κανονισμό Eurodac. Πέμπτο στοιχείο του πακέτου, το αναθεωρημένο επιχειρησιακό σχέδιο της ε, κοινή επιχείρηση τρίτων. Το συζητούμε εδώ και 12 μήνες από όταν πρώτο εμφανίστηκα στην Επιτροπή σας. Εσείς πιέζετε ε, έντονα προκειμένου να εστιάσουμε στην ε, σωτηρία ε, ζωών Γιατί και τα τελευταία πολύ δυσάρεστα γεγονότα του Απριλίου έδωσαν μια πολιτική όθηση για την ε, διεύρυνση της ε, επιχείρησης τρίτων. Ε, διευρύνεται λοιπόν η γεωγραφική κάλυψη του τρίτων προς νότον αναπτύσσονται περισσότερα μέσα ε, αυξάνεται ο προπολογισμό, χάρη σε εσά και στη βοήθειά σας βέβαια και να σας δώσω ένα εντυπωσιακό στοιχείο. Από την 1η Μαΐου και μέχρι τις 30 ε, Ιουνίου σε 300 περίπου επεισόδια Είχαμε 269 περιπτώσεις ε, έρευνας και εντοπίσαμε πάνω από 44.000 άτομα και διασώσαμε 33.855 άτομα, άντρες, γυναίκες και παιδιά. Μόνο δύο διαπιστωμένους θανάτους καταγράψαμε. Ε, σημαντική αλλαγή για την οποία μπορείτε και εσείς να είστε περήφανοι εδώ στην Επιτροπή σας, διότι πάντοτε ε, μάχεστε ε, υπέρ των επιχειρήσεων διάσωσης. Τέλος, για να σας δείξω πόσο ολιστική είναι η προσέγγιση μας, θελήσαμε να συμπεριλάβουμε και ένα και στοιχείο νόμιμης μετανάστευσης στο θεματολόγιο. Γι' αυτό το λόγο ξεκινήσαμε διαβούλευση για το θέμα της μπλε κάρτας, της αναθεώρησης του συστήματος μπλε κάρτας. Η δημόσια αυτή διαβούλευση ξεκίνησε πριν από μερικές εβδομάδες. Τα αποτελέσματα θα μας δείξουν το δρόμο για την αναθεώρηση του συστήματος μπλε κάρτας. Η διαβούλευση εξακολουθεί να είναι ανοιχτή για 12 εβδομάδες μέχρι τέλος Αυγούστου, 22 Αυγούστου πιο συγκεκριμένα. Θα ήθελα να σας ζητήσω να την κάνετε γνωστή αυτή τη διαβούλευση έτσι ώστε να πάρουμε όσο το δυνατό περισσότερες απαντήσεις γίνεται. Ευχαριστώ. Thank you very much, um, uh, Ευχαριστώ Ματίας. Υπάρχει αυτή τη βδομάδα ένα συμβούλιο Τζάι, mm. όπως αναφέρθηκε από τον συνάδελφο, και ελπίζουμε ότι στο θέμα της μετεγκατάστασης, του μηχανισμού μετεγκατάστασης θα υπάρξει πρόοδος. Η Σκάρ Κέλλερ είναι η συγγήτρια για τη διαβούλευση και πώς θα συζητήσουμε λοιπόν πριν ακούσω τους ευρωβουλευτές. Θα ήθελα η Λουξεμβουργιακή Προεδρία, συντομία, ε, να μας μιλήσει. Ελπίζω ήδη αυτή την εβδομάδα να προχωρήσουν τα πράγματα. Η Σκά θα είναι παρούσα. Αν μπορούσε λοιπόν η Προεδρία πολύ σύντομα να μας πει τι περιμένουμε αυτή τη βδομάδα να δούμε. Ε, και εν συνεχεία η ΣΚΑ Κέλλερ θα μας κάνει μια σύντομη παρουσίαση. Ο κ. Κιέγγε για την στρατηγική έκθεση επίσης και άλλος ένας συνάδελφος θα κάνουν μια σύντομη εισαγωγή και εν συνεχεία θα ακούσουμε τις ερωτήσεις. Παρακαλώ λακωνικά γιατί καταλαβαίνετε ότι έχουμε ένα πολύ μακρύ κατάλογο από μιλητές. Και φυσικά να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι έχουμε και δύο εξωτερικούς ομιλητές οι οποίοι προέρχονται από δύο οργανώσει πλειοκτητών. Ε, θα είναι πολύ ενδιαφέρον να του ακούσουμε. Καλό να του δώσουμε λοιπόν τον απαραίτητο χρόνο. Να ακούσουμε λοιπόν καταρχήν τη Λουξεμβουργέζικη Προεδρία να μας πει το, τα σχέδιά τη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επιτρέψτε στην Προεδρία να πει δύο λόγια για την ατζέντα σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση και πιο συγκεκριμένα για την απόφαση σε ό,τι αφορά τη κατάσταση η Κομισιόν ε, καθόρισε την ατζέντα της που είναι η βάση εργασίας μας ε, για το θέμα αυτό. Οι διαβουλεύσεις ε, υπό την αιγίδα της Προεδρίας δείχνουν ότι πρέπει να προβληματιστούμε εντελεχώς για την πολιτική τη Ευρώπη για τη μετανάστευση. Η κατάσταση επιτόπου μα αναγκάζει να επιταχύνουμε τη διαδικασία μεταρρυθμίσεων. Ω Προεδρία του Συμβουλίου θα ασχοληθούμε με το καθήκον αυτό με την υποστήριξη των κρατών μελών. Θα πρέπει να προωθήσουμε ε, σφαιρικά το θέμα αυτό δεν θα πρέπει να υπάρχουν ε, στρεβλώ ό,τι αφορά τι μεταναστευτικέ ροέ. Θα πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη σε ό,τι αφορά την προσπάθεια που θα κάνουμε όλοι, σε ό,τι αφορά την κοινωνική βοήθεια, είτε οικονομική, είτε μέσω των εξειδικευμένων φορέων και οργανισμών. Θα προχωρήσουμε με αραγέ μέτωπο, ε, με μια λογική πακέτου. Ε, ευθύνη, αλληλεγγύη, νόμιμη εισαγωγή και συνεργασία διεθνής. Ο σημερινό σχεδιασμό προβλέπει τουλάχιστον τρει μεγάλε πολιτικέ συζητήσει σε επίπεδο Συμβουλίου Τζάι. Ε, αυτή τη βδομάδα είπατε, ε, στη συνεδρία στην Άτυπη, θα γίνει μια συζήτηση για το σχέδιο δράση ε, μετανάστευση για την επανεκατάσταση και την μετεγκατάσταση. Τον Οκτώβριο θα γίνει μια συζήτηση για την ανάπτυξη τη θεωρήση και την πολιτική επιστροφών και το Δεκέμβριο το μέλλον των εξωτερικών συνόρων. Μια συνέχιση για όλε τι δράσει θα σε επίπεδο hot spot ε, με τους αξιωματικούς συνδέσμους, ε, την εφαρμογή της Eurodac, το, το κέντρο στον Ήγυρα ε, και τα θέματα της επανειστοχής και των επιστροφών. Στο Στη Σύνοδο Κορυφή η Προεδρία προτείνει να προχωρήσουμε γρήγορα με βάση ένα κατάλογο σίγουρων χωρών για το διεθνέ πλαίσιο. Η Σύνοδο Κορυφή τη Βαλέτα έχουμε γι' αυτό μια ειδική ομάδα με στόχο να κάνουμε μια πολιτική δήλωση και να δούμε ποιε είναι οι δράσει προτεραιότητα μαζί με του ε, ε, Αφρικανού εταίρου. Η Υπουργική Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου για τον, ε, την οδό των Βαλκανίων. το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επικύρωσε τι αρχέ και οι προβληματισμοί έχουν ξεκινήσει πάνω σε αυτό το θέμα. Επιπλέον, η Προεδρία δεσμεύεται να συνεργαστεί και να δουλέψει πάνω σε φακέλους όπου ε, ερευνητές, φοιτητές, ε, ασυνόδευτοι ανήλικοι. Δεν χρειάζεται να διευκρινίσω στον χώρο αυτό ότι πραγματικά θέλουμε να τελεσφορήσουμε σε αυτά τα θέματα. Επιτρέψτε μου επίσης ε, καταληκτικά να πω δύο λόγια για το θέμα της επανεκατάστασης και μετεγκατάστασης. Όλοι διαβάσατε τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπω σε λεπτομέρειες για ό,τι λένε. Ξέρετε ότι σε ό,τι αφορά πιο συγκεκριμένα την απόφαση του Συμβουλίου για προσωρινά μέτρα σε ό,τι αφορά την μετεγκατάσταση. Οι εργασίε είναι εξελίξη και η πρώτη ομάδα εργασία ε, έγινε συνεδρία την περασμένη εβδομάδα. Το Κορεπέρα ασχολήθηκε σε μια συνεδρίαση που ασχολήθηκε αποκλειστικά με αυτό το θέμα σήμερα το πρωί και άλλε συνεδριάσει θα ακολουθήσουν αυτή τη βδομάδα και τι επόμενε εβδομάδε. Μεταξύ των θεμάτων που είναι σήμερα αντικείμενο συζήτηση, μπορώ να φέρω μεταξύ άλλων την αξιολόγηση, την τακτική των ομάδων δικαιούχων, ε, δευτερογενή κινήματα, ε, επιχειρησιακή βοήθεια στην Ιταλία και στην Ελλάδα, καθώ και θέματα που αφορούν την ε, ένταξη των ενδιαφερομένων αυτών ατόμων. Σε ό,τι αφορά τα νούμερα και τις δεσμεύσει. Τα νούμερα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι ξεκάθαρα. Η η Προεδρία ξεκίνησε τις διαβουλεύσεις και είναι εξελίξη, θα συνεχιστούν. Δουλεύουμε πολύ αποφασιστικά για να έχουμε ένα αποτέλεσμα μέχρι το τέλος Ιουλίου και θα είναι ένα σημαντικό βήμα το άτυπο συμβούλιο αυτής της εβδομάδας όπου ο πρόεδρος Μόρες, ε, ο Λουξεμβουργίας δηλαδή πρόεδρος, θα συμμετάσχει. Ευχαριστώ. Okay, thank you very much. Um, Ευχαριστώ πολύ. Σκάκελα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Επιτροπή και την Προεδρία που ήρθε, έκανε την παρουσίαση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έκανε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση νομίζω και όλοι βλέπουμε τα αποτελέσματα. Και από την πλευρά μου το απογοητευτικό ήταν ότι επί ενός συμβολικού μέτρου όπου όλοι θέλουμε συμφωνία επί ενός ευρωπαϊκού α, μηχανισμού αλληλεγγύης ένα κράτος μέλος δεν συμμετείχε. Η αλληλεγγύη ήταν σε θελοντική βάση, αλλά η αλληλεγγύη δεν ξέρω πώς μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη. Με τις εκθέσεις του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ κυρίως μπορεί να στείλει σαφές μήνυμα στα κράτη-μέλη. Δυστυχώς θα μας διαβουλευθούν για τον μηχανισμό ε, επίγουσας ανάγκης. Θα επανέλθω σε αυτό. Πάντως είναι πολύ σημαντικό να αποστείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα και να ζητήσουμε δεσμευτικό μηχανισμό. Αυτό έχει γίνει ήδη σε ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στις 28 Απριλίου του 2015 όπου ζητήσαμε δεσμευτική ποσόστοση για τη διανομή των ετούντων άσυλων σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό πρέπει να το ξαναπούμε ξανά και ξανά και εμείς στο Κοινοβούλιο να αποστείλουμε ηχηρό μήνυμα ότι θέλουμε δεσμευτικό μηχανισμό ώστε να ε, είναι αποτελεσματική η αλληλεγγύη στην πράξη. Αναφέρθηκαν ε, οι στόχοι των 40.000 από την Κομισιόν θα έλεγα ότι τα κράτη-μέλη δεσμεύτηκαν να αναλάβουν 40.000 ετούντες άσυλο από την Ιταλία και την Ελλάδα και η Κομισιόν σε αυτό το νούμερο έλαβε μόνο υπόψη τα στοιχεία από το 2014. Όμως, αν δούμε τα νούμερα που είχαμε τους πρώτους μήνες τρέχοντος έτους, βλέπουμε ότι τα νούμερα αυξάνονται. Τους πρώτους μήνες του 2015 έρχονται πολύ περισσότεροι από ότι την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Γι' αυτό νομίζω ότι το μήνυμα που μπορούμε να στείλουμε είναι ότι δεν σταματάμε στους 40.000, αλλά θα πάρουμε αρχικά το στοιχείο αυτό, τον αριθμό αυτό της ε, Κομισιόν, αλλά θα το επεκτείνουμε το 2015 και καταλήγω έτσι ότι ο στόχος μας πρέπει να είναι 50.000 ετούντες άσυλο που πρέπει να ε, μετεγκατασταθούν από την Ιταλία και την Ελλάδα. Να σας δώσω και ένα αριθμητικό στοιχείο. Στην Ελλάδα οι αφήξεις εξαπλασιάστηκαν σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι. Οπότε τώρα έχουμε, και τώρα έχουμε πολύ περισσότερες ε, αφήξεις στην Ελλάδα από την Ιταλία. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να στείλουμε ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης. Ας είναι συμβολικό να πούμε ότι χρειάζεται περισσότερη αλληλεγγύη με τρόπο δεσμευτικό και μην ξεχάσουμε να θέσουμε υψηλούς στόχους. Πρέπει όμως να δούμε και την ποιότητα του μηχανισμού, όχι μόνο να δούμε ποσοτικά το θέμα των θέσεων που θα προσφέρουμε. Είχαμε ένα παράδειγμα ήδη όπου ένα έγινε με την εγκατάσταση στα πλαίσια του Γιουρίμα, πιλωτικό πρόγραμμα πριν από λίγο καιρό στη Μάλτα. Και κάποια διδάγματα πρέπει να αντλήσουμε από αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα στην Μάλτα. Δεν ήταν πολύ καλή η εμπειρία, η Μαλτέζικη, και αυτό έχει να κάνει και με τους ίδιους τους μετανάστες που αντιμετωπίστηκαν ως νούμερα. Αριθμούς που μπορούσαν να τους πηγαίνουν παραπέρα χωρίς διαβουλεύσεις άλλα κράτη-μέλη. Είχαμε πολλές ε, δεύτερο γενείς μετακινήσεις μετά. Τα κράτη-μέλη συμφωνούν νομίζω ότι καλύτερα είναι να αποφεύγονται αυτές οι δευτερογενείς μετακινήσεις. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Αλλά πώς να επιτευχθεί. Νομίζω ότι θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε εκεί που υπάρχει κάποια προτίμηση από την πλευρά του ετούντος, διότι έχει συγγενείς, διότι είναι η γλώσσα ε, πρόσφορη, ή έχει σχέσεις, επαφές, ή έχει μια κοινότητα ε, συμπατριωτών. Αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Και βέβαια δεν πρέπει να τα κάνουμε όλα ε, πάντοτε υπόψη, δεν είναι δεσμευτικό αυτό, αλλά Όπου μπορούμε, καλό είναι οι προτιμήσεις να λαμβάνονται υπόψη, ούτω ώστε να διευκολύνουμε τους ανθρώπους να εντάσσονται, να ενσωματώνονται στην ε, δεύτερη τους χώρα και να βελτιώνονται. Να βλέπουμε και τις προτιμήσεις των κρατών μελών επίσης, γιατί αν συντεριάζονται οι, προτιμήσει, προτιμήσεις, τότε έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα, γιατί και θα ενταχθούν και θα μείνουν εκεί που τους στείλαμε θα έχουν καταλάβει δηλαδή γιατί έφτασαν εκεί και θα μείνουν εκεί. Ενώ αν ε, δεν καταλαβαίνουν δεν μπορούν να ενσωματωθούν. Αυτό είναι σημαντικό. Είναι ένα δίδαγμα που άγγισε από το πρόγραμμα Γιουρίμα. Πρέπει λοιπόν να διευκολύνουμε με αυτόν τον τρόπο την επιτυχία του προγράμματος και νομίζω ότι πρέπει να πετύχει ώστε να έχουμε και άλλους μηχανισμούς αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών που θα μπουν σε λειτουργία. Είναι λοιπόν και αυτό το ποιοτικό στοιχείο πολύ σημαντικό. Και συνεχίζω. Ήδη σας είπα για το κατεπήγον αυτό μέτρο που είναι λίγο περίεργο για το Κοινοβούλιο γιατί επειδή είναι κατεπήγον, είναι μέτρο επίγουσας ανάγκη, γίνονται μόνο διαβουλεύσεις με το Κοινοβούλιο δεν ε, είναι συνομοθέτης όπως θα έπρεπε το Κοινοβούλιο προκειμένου. Πρέπει να τονίσουμε λοιπόν ότι μπορεί να δεχτεί αυτές τις διαβουλεύσεις στο Κοινοβούλιο γιατί είναι μηχανισμός επίγουσας ανάγκης και μόνο σε αυτή την περίπτωση η Κομισιόν ε, θα δράσει έτσι. Όμως μας υποσχέθηκε μέχρι το τέλος του χρόνου να μας δώσει ε, ένα πιο μόνιμο πρόγραμμα και εκεί βέβαια θα παίξει το συνήθι ρόλο του το Κοινοβούλιο συνομοθέτης. Να τονίσουμε όμως ότι αυτό πρέπει να το δούμε. Και αν η Κομισιόν δεν αντιδράσει σε έφθετο χρόνο τότε το Κοινοβούλιο ε, θα σκεφτεί την δυνατότητα να συντάξει δική του έκθεση πρωτοβουλίας. Γιατί το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να διαβουλεύεται μόνο ε, ως νομοθέτης, πρέπει να παίξει το ρόλο του, το νομοθετικό. Αυτές είναι οι βασικές γραμμές της έκθεσης. Όλοι οι σκιώδεις είδαν την, το πλήρες κείμενο. Προσβλέπω στα σχόλιά σας, στις προτάσεις σας. Δυστυχώς είναι πολύ μικρή η προθεσμία. Ε, ήταν πολύ φορτωμένο το πρόγραμμα του Συμβουλίου. Πρέπει όμως να αρχίσει ο μηχανισμός με την κατάσταση relocation να τεθεί γρήγορα σε λειτουργία. Τέλος να, να ευχαριστήσω τους βοηθούς και τους συμβούλους και τη γραμματεία όλοι βοήθησαν, αλλιώς δεν θα προλαβαίναμε. Και δουλέψαμε σε χρόνους ρεκόρ για να ετοιμαστεί η έκθεση. Ευχαριστώ για τη συνεργασία που το κατέστησε αυτό δυνατό. Ευχαριστώ. να προσθέσω και εγώ κάτι σε αυτά που είπε. Καταρχά ε, σα ευχαριστώ που ήρθατε όλοι δευτεριάτικα στο Στρασβούργο. Αν δεν είχαμε κάνει σήμερα το βράδυ αυτή τη συνεδρίαση, δεν θα μπορούσαμε να σεβαστούμε το χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ λοιπόν του συναδέλφου για την ευελιξία του να παραστούν Δευτέρα βράδυ στο Στρασβούργο. Τώρα, οι συνάδελφοι, ακούσαμε την ε, εισηγήτρια, ακούσαμε την Προεδρία και την Κομισιόν και τώρα θα ακούσουμε με του Ευρωβουλευτέ τους συζητητέ ε, με εκθέσει ε, ιδίας πρωτοβουλία. Η Ρομπέρτα δεν μπορούσε να έρθει. Ο Γερούν όμως ε, θα πάρει τη θέση της και θα πει δύο λόγια εκ μέρου της. Παρακαλώ συνάδελφοι, εάν μπορείτε να μην ξεπεράσετε τα δύο λεφτά, καλό θα ήταν γιατί έχουμε ένα το κατάλογο ομιλητών. Γύρω στα δύο λεφτά αν μπορείτε. Η παρουσίαση της έκθεσης Ε, έχουμε και την έκθεση για τη διαβούλευση που έγινε για, το, για τη μετεγκατάσταση. Ήταν λογικό που τη δώσαν 5-6 λεπτά. Η Ρομπέρτα. Ε, προσπαθεί ακόμα να φτάσει στο Στρασβούργο. Ελπίζω ότι θα φτάσει κάποια στιγμή έγκαιρα, έτσι ώστε να ακούσουμε και από το δικό τη στόμα τι απόψει τη. Ε, σίγουρα πολύ πιο γλαφυρά από ότι θα το κάνω εγώ σε ό,τι αφορά τον, το θέμα του μηχανισμού μετεγκατάστασης. Πρόκειται για μια ευκαιρία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συμφωνώ με την Σκάκελερ ότι το αποτέλεσμα της συνεδρίας του Συμβουλίου ήταν απογοητευτικό και η ατμόσφαιρα στην οποία έλαβαν χώρε συζητήσει, σύμφωνα με τα όσα διάβασα στον τύπο, ε, δεν, ήταν, δεν μας κάνει καθόλου περήφανους. Οπότε συμφωνώ με την εισηγήτρια και τους και εισηγητές. Ε, θα πρέπει η Ευρώπη να δείξει πιο ενωτική συμπεριφορά και να δώσει στους πολίτες αυτό που περιμένουν από εμά. Σε ό,τι αφορά το πακέτο αυτό, χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το υπέβαλε. Παρ' όλα αυτά πρόκειται για μία από τις προτάσεις του θεματολογίου. Προκειμένου να λειτουργήσει όλο το θεματολόγιο πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή και να υλοποιηθούν όλα τα πακέτα, τα εφαρμοστικά πακέτα. Θα πρέπει να ε, αντιμετωπίσουμε τις, ε, τα δίκτυα, να ακολουθήσουμε ε, αποτελεσματικές στρατηγικές επιστροφής, ε, να δούμε τις σχέσεις με τον Ήγηρα, όλα αυτά πρέπει να συνοδεύσουν το πακέτο το οποίο μας υποβλήθηκε. Τι μπορούμε να προσθέσουμε εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρώτον, η ιδέα του να λαμβάνονται υπόψη οι προτιμήσεις των ε, μεταναστών. Υπό το φως ιδιαίτερα της εμπειρίας της Μάλτας. Παρ' όλα αυτά, οι προτιμήσεις αυτές μπορούν να ληφθούν υπόψη μόνο στο μέτρο του δυνατού. Δεν νομίζω ότι οι μετανάστες θα έχουν ένα μενού από το οποίο να μπορούν να διαλέξουν. Αν μπορέσουμε όμως να ικανοποιήσουμε ορισμένες αυτές τις προτιμήσεις, ακόμα καλύτερα. Αυτή η ιδέα βέβαια δεν θα πρέπει να προσθέσει πολύ γραφειοκρατία. Δεν θα πρέπει να προσθέσει πολύ διοικητικό άχθος προκειμένου η προστασία σε όσους τη χρειάζονται να δίδεται το συντομότερο δυνατό, αποφεύγοντας την υπέρμετη γραφειοκρατία. Επίση, είναι σαφέ ότι αυτό αποτελεί, αυτό το, η πρόταση είναι κάτι σαν πιλωτικό πρόγραμμα και η Κομισιόν επεξεργάζεται ένα μόνιμο μηχανισμό έκτακτης ανάγκη, παρόλο που αυτό δείχνει αντιφατικό, έτσι, ε, μόνιμο και ε, έκτακτο στην ίδια φράση. Ε, περιμένουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρόλα αυτά θα έχει εξουσία στην απόφαση σε σχέση με αυτό το μόνιμο πακέτο, το μόνιμο μηχανισμό. Και είναι σημαντικό, ακόμα σημαντικότερο, να πετύχει αυτό το πρώτο πιλωτικό σύστημα. Εγώ είμαι υπέρ ενό υποχρεωτικού συστήματος ε, κατανομής ε, ε, μετεγκατάσταση, αλλά δεν νομίζω ότι είναι η στιγμή αυτή πιο κατάλληλη για να συζητήσουμε τα νούμερα της πρότασης. Είναι πολύ πιο σημαντικό να πειραματιστούμε με το μηχανισμό, να δούμε πώς λειτουργεί και να διαπιστώσουμε πώς μπορεί να βελτιωθεί. Όλα αυτά να τα λάβουμε υπόψη όταν συζητήσουμε τον μόνιμο μηχανισμό. Οπότε, ανυπομονώ να συνεργαστώ με την εισηγήτρια και τους ε, σκιοσηγητές. Ε, στο τελευταίο χρόνο, τον πρώτο μου χρόνο στο Κοινοβούλιο, δεν έχω δει τόσο αποτελεσματική εργασία ως τώρα. Οπότε, συγχαρητήρια, ευχαριστώ. as well as nominated by uh, Είσαστε και εκπρόσωπος της κυρίας Μετσόλα και μιλάτε και ως ε, σκιώδης συγητής. Είσαι σύλλη τώρα. Θα μιλήσει για την έκθεση Δίας Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την δουλειά της και για τις τροπολογίες που επέφερε στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου. Η εισηγήτρια έκανε προτάσεις πολύ σημαντικές. Ξεκινώντας καταρχήν από την ενίσχυση της ε, υποχρεωτικότητας των ποσοστώσεων κατανομής. Ακόμα και η νέα διάταξη για τη δυνατότητα που παραχωρείται στον μετανάστη να εκφράσει μια προτίμηση για τη χώρα υποδοχής του είναι σημαντικό. Έχω κάποια επίκριση σε ό,τι αφορά την αύξηση των αριθμών των μεταναστών που θα μετεγκατασταθούν σε ευρωπαϊκό έδαφος. Κατά την άποψή μου, όπως είπε και η συγγήτρια, καλύτερο θα ήταν να επιμείνουμε είτε για ένα σημαντικό αριθμό ε, μεταναστών που μετεγκαθίστατο ή να μιλήσουμε για ένα αξιόπιστο ποσοστό, ούτω ώστε να ε, πάρουμε από τους ώμου κάποιων κρατών μελών το βάρος. Συμφωνώ με την συγγήτρια που μιλάει για την ε, νομική βάση. Ε, το άρθρο 78.3 το μεταναστευτικό φαινόμενο δεν έχει πάντα ε, επίγοντα χαρακτήρα. Μερικές φορές έχει διαρθωτικό χαρακτήρα, εξού και η κριτική. Γι' αυτό λοιπόν θα μπορούσαμε ε, να έχουμε άλλες νομικές βάσεις. Το 78.2 και το άρθρο 80 για τις επακόλουθες πράξεις. Σε ό,τι αφορά τη δουλειά που κάνουμε με τη συνάδελφό μου Ρομπέρτα οι προπαρασκευτικές εργασίες για τα έγγραφα εργασίας που θα οδηγήσουν στη σύνταξη της έκθεσης πρωτοβουλίας ε, ετοιμάζονται. Ε, ίσως έχουμε καθυστερήσει σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που είχαμε καθορίσει, αλλά συνολικά δεν θα καθυστερήσουμε. Δεν θα... Με κοινή πρωτοβουλία ε, θεωρήσαμε ότι είναι σημαντικό να κάνουμε μια συζήτηση αφού μιλήσαμε όλους τους συναδέλφους της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και τους μοιράσαμε τα έγγραφα εργασίας, ούτως ώστε να τους ενημερώσουμε για να μπορέσουν να παρουσιάσουν πιο συγκεκριμένους προβληματισμούς. Επίσης, αναβάλαμε τη συνάντηση που θα είχαμε σήμερα για τις νόμιμες οδούς ε, ή ασφαλείς οδούς πρόσβασης, ούτως ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε με τους κοιόδης συζητητές. Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο για να δουλέψουμε επί ενός κειμένου που θα συμμεριζόμαστε όλοι. Θέλω να πω δύο λόγια, να ευχαριστήσω τον Διευθυντή των πλειοκτητών, της Οργάνωσης Πλειοκτητών για τη συνεισφορά του. Τις περασμένες ημέρες είχαμε μια συνάντηση με την οργάνωση αυτή των εφοπλιστών για να δούμε ε, τι δράσεις προωθούν και αυτοί. Όπως υπόθηκε, θεωρώ ότι οι σωστικές ε, ενέργειε δεν μπορούν να αφαιθούν μόνο σε ιδιώτε. Είναι ευθύνη των κρατών μελών να δώσουν τα, μέτρα, τα μέσα και τη χρηματοδότηση για να εξασφαλίσουν τις ε, ε, σωστικές δραστηριότητες με επαγγελματικότητα και με συγκεκριμένα κριτήρια. Αφού άκουσα την παρουσίαση των μέτρων για την του θεματολογίου της μετανάστευσης θα ήθελα να σταθώ σε κάποια σημεία. Μέχρι τώρα στην Ευρώπη Υπάρχει ένα κλείσιμο σε ό,τι αφορά την νόμιμη μετανάστευση για λόγους ε, οικονομικούς. Η Κομισιόν με τις δικές της προτάσεις δεν πρότεινε ε, καλές λύσεις. Νομίζω ότι θα πρέπει να δουλέψουμε πολύ από αυτού του θέματος. Να παρέμβουμε στις πραγματικές αιτίες ε, της μετανάστευσης και της μετακίνησης ε, των ανθρώπων αυτών. Η κατάσταση στη χώρα από την οποία φεύγουν αυτά τα άτομα και οι νόμιμες οδοί άφηξη στην Ευρώπη για άτομα τα οποία χρήζουν διεθνού προστασία και για τους πρόσφυγες. Κλείνοντα, θα ήθελα να ζητήσω από το Διευθυντή να μου απαντήσει ένα ερώτημα. Ε, εσχάτως ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με τον επαναπατρισμό. Ε, υπό την αιγύρια του Συμβουλίου η συζήτηση αντί να σταθεί στην αλληλεγγύη μιλάει κυρίως για κατασταλτικά μέτρα. Χωρίς διακρίσεις. Επανα, ε, επαναπατρισμός. Εμείς θα θέλαμε καμία πολιτική επιστροφής να μην ε, προωθείται με τρόπο αφαίρετο, χωρίς ε, από απόλυτου σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισχύουσας νομοθεσίας. Γι' αυτό ζητάω από την Κομισιόν. Αν έχετε πάρει προληπτικά μέτρα για να εμποδίσετε κάποια κράτη-μέλη να, βάλουν, να επιβάλλουν πολιτικές ε, επαναπατρισμού που περιορίζουν τις ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ευχαριστώ. okay. Ωραία. Ωραία. Έχετε υπόψη και το χρόνο. Είναι μεγάλος ο κατάλογος ομιλητών. Και επικεντρωθείτε στην, στο μηχανισμό μεταγκατάστασης, γιατί αυτό θα συζητηθεί στο Συμβούλιο αυτή την εβδομάδα. Και όπως είπε και η Σκά Κέλλερ, εμείς θέλουμε να παρουσιάσουμε τις δικές μας απόψεις την Πέμπτη στο Συμβούλιο στους Υπουργούς. Είναι σημαντικό να πούμε τι πιστεύουμε για το μηχανισμό στο Συμβούλιο Τζάι. Η κυρία Χολμάιερ. Δύο βασικά ερωτήματα στον κύριο Ρούτε. Πρώτη ερώτηση. Πιστεύετε ότι ανάλογα με το πώς αποφάσισαν οι αρχηγοί των κυβερνήσεων κάποια στιγμή υπάρχει ενδεχομένως να έχουμε ε, έναν μηχανισμό κρίσεων που θα έχει εξομαλυνθεί και θα λειτουργεί χωρίς να επικεντρώνεται σε συγκεκριμένο αριθμό αλλά θα ενεργοποιείται όταν ένα κράτος μέλος έχει να αντιμετωπίσει ε, πολύ μεγάλους αριθμούς μεταναστών προσφύγων και δεν μπορεί να ανταποκριθεί μόνο του. Δεύτερη ερώτηση. Ο Επίτροπος Αβραμόπουλος ε, μίλησε για ένα, μια αιστεία προβλήματος στην Σικελία για την Ουγγαρία. Χαίρομαι που θα δημιουργήσει ένα hot, θα, θα αντιμετωπιστούν αυτά τα hot spots, αλλά πώς συγκεκριμένα, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κατάσταση από το ένα hot spot στο άλλο, έτσι χωρίς άλλο χρειάζεται προσωπικό, χρειάζεται χρειάζονται προϋποθέσεις λειτουργίας και καλή συνεργασία με το κράτος, κράτος μέλος. Βέβαια, ε, αυτές είναι ερωτήσεις προς τον κύριο Ρουίτε που θα απαντήσει στο τέλος της συνεδρίασης. Η Μπέργκητ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, ίσως είναι προφανές αλλά έχοντας υπόψη μας ε, κάποιες συζητήσεις δημόσιες, δημοσιευμένες, εκτιμώ ότι ο κ. Σουρίτε είπε ξανά με πολύ ξεκάθαρο τρόπο αυτήν την ολιστική προσέγγιση ε, στη μετανάστευση. Δεν μπορούμε δηλαδή να ε, μιλήσουμε για ένα μέτρο μόνο, αλλά θα υπάρξει πρόοδος στο θέμα μετανάστευση αν λάβουμε υπόψη μας όλα τα θέματα με την κατάσταση περιορισμού της λαθρέας διακίνησης ε, και όλα αυτά πρέπει να τα κάνουμε ταυτόχρονα και με μεγάλο ε, ζήλο για να έχουμε αποτελέσματα. Χαίρομαι που το είπατε αυτό. Ερώτηση τώρα. Όταν αρχίσατε να μιλάτε για την Ελλάδα, αν σας κατάλαβα καλά, είπατε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα γιατί οι πρόσφυγες τώρα δεν έρχονται από τα χερσαία σύνορα αλλά μέσω θαλάσσης ε, και έτσι είναι πολύ δύσκολο να έχουμε ε, συγκεντρωπημένο συγκεντρωτικό σύστημα για να αντιμετωπίσουμε πολλά τα νησιά. Ίσως είναι παράδοξο το ε, ερώτημα, αλλά ίσως αυτό θα διευκόλυνε να ανοίξετε σε ένα σημείο το φράχτη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ώστε οι πρόσφυγες να περάσουν από εκεί, από αυτό το πέρασμα και να υπάρχει ένα κεντρικό σημείο υποδοχής και όχι ε, διάφορα διάσπαρτα στην περιοχή. Επίσης, για την οικονομική υποστήριξη, 6.000 ευρώ για τη μετεγκατάσταση είπαμε. Ξέρουμε ότι είναι διαφορετικά τα κέντρα. Δηλαδή, οι 6.000 ευρώ στη μια χώρα μπορεί να είναι πολλά. Σε μια άλλη χώρα μπορεί να μην είναι τίποτα. Παράλληλα, εδώ μεταξύ, κάποια κράτη-μέλη ήδη είναι λίγο πολύ καλά προετοιμασμένα για να αντιμετωπίσουν τη μετανάστευση, ενώ άλλα όχι. Δεν πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν άλλον μηχανισμό για να αποφασίσουμε αν και σε ποιο βαθμό τα κράτη-μέλη μπορεί να χρειάζονται πρόσθετα κονδύλια. Άλλη ερώτηση. Ως πρόσθετο στοιχείο στην κλίδα κατανομής μπορούμε ίσως να λάβουμε υπόψη μας κάποιες επιθυμίες των προσφύγων. Στο βαθμό που είναι σαφές ότι στο τέλος μπορεί να μην ε, μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις επιθυμίες, συμφωνώ. Να πούμε δηλαδή αν έχετε μία, δύο, τρεις ε, χώρες που προτιμάτε γιατί έχετε συγγενείς εκεί κλπ. Καλό είναι αυτό το σημείο εκκινήσεως για να νιώσουν και εκείνοι κάπως πιο ε, εύκολα. Για τον αριθμό των μετεγκαταστάσεων, ναι, σε σχέση με άλλες χώρες γύρω από την Ευρώπη, ο αριθμός των 40.000 προσφύγων και η συνολική αριθμή που έχουμε εδώ Πράγματι είναι γελία μεγέθη, γιατί πολλές χώρες έχουν υποδεχτεί, αναλάβει περισσότερους πρόσφυγες από ότι εμείς στην Ευρώπη. Οπότε ο αριθμός των 40.000 δεν φαίνεται μόνο, αλλά είναι όντως κάπως ε, αστείος. Από την άλλη πλευρά όμως για να είμαστε ειλικρινείς αν μπορούμε να αρχίσουμε με τις 40.000 και αν όλα τα κράτη-μέλη συμμετάσχουν, αυτό είναι καλό. Δηλαδή, να σταματήσουν να λένε ότι έχουν διαφορετικά προβλήματα, γιατί κάθε, όλα τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικά προβλήματα. Εγώ όμως θέλω να κάνουμε μια αρχή, να γίνει αυτή η ανταλλαγή ε, πρακτικών και να δουλέψουμε πάνω στα προβλήματα που έχουμε. Η Ευρώπη είναι θεμελιωμένη σε κάποιες αξίες, κοινέ αρχές και θα τις κρατήσει ακόμα και σε περίοδο ισχνών αγελάδων και αντικσοοτήτων. Εντάξει, από ό,τι φαίνεται δεν προεδρεύω πολύ καλά γιατί με αγνοείτε. Ε, και αυτά τα δύο μαζί φέρνουν καταστροφή. Τρίτον, υπάρχει και άλλο ένα κατάλογο ομιλητών, τον οποίο δεν είχα δει. Όλα αυτά μπορώ να τα περιγράψω μόνο ως κόλαση. Τέταρτον, έχουμε και προσκαλισμένους ομιλητές. Οπότε, Τώρα περιορίζεται ο χρόνος αγόρευσης σε 1,5 έως 2 λεπτά. Παρακαλώ πολύ λάβετε το υπόψη σα. Γιατί θα σα διακόπτω. Σας παρακαλώ πολύ λοιπόν προσπαθείτε Προσπαθήστε να περιοριστείτε στο 1,5 με 2 λεπτά. Σεσίλια, ευχαριστώ πολύ την Κομισιόν για την παρουσίαση και την προσήλωσή της. Ε, δεδομένης όμως η κατάσταση στο Συμβούλιο, αμφιβάλλω αν θα καταφέρουμε να ε, εγκρίνουμε κάποιο υποχρεωτική εφαρμογή σύστημα. Και αυτή είναι η ερώτηση η Κομισιόν θα μπορούσε να δεχθεί ένα τέτοιο σύστημα εθελοντικά ή αλλιώς πώς θα μπορούσαμε να διασφαλίσουμε ότι όλα τα κράτη-μέλη θα λάβουν τις ευθύνες τους και θα συμμετάσχουν. Εγώ πραγματικά έχω βαρεθεί. Ε, με εκνευρίζει που βλέπω ότι υπάρχουν κράτη-μέλη που μιλούν για τη δημιουργία, για το χτίσιμο τείχων στην Ευρώπη και δεν θέλουν να πάρουν τυχόν μάλλον να το πούμε έτσι στην Ευρώπη και δεν θέλουν να δεχθούν ούτε ένα ετούντα άσυλο. Ε, ή έχουμε ευρωπαϊκή ελεγγύη ή όχι. Ξέρουμε τι συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα. Εδώ θα πρέπει να δείξουμε την αλληλεγγύη μας και, σε ένα, και στο επόμενο μάλιστα επίπεδο. Είναι πολύ σημαντικό. Είμαι υπέρ των παρατηρήσεων της Κακέλερ. Η πρόταση είναι πολύ φιλόδοξη και ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να είμαστε και εμείς φιλόδοξοι στις υποσχέσεις μας, στις δεσμεύσεις μας. Θα πρέπει να πιέσουμε τα κράτη-μέλη να καταλάβουν και να αναλάβουν την ευθύνη του το καθένα. Ευχαριστώ. Σαφέστατο. Μόνο... Η Κορνίλια. Ευχαριστώ. Μιλήσατε για το Δουβλίνο, ότι είχε επιτυχία. Όχι. Καθόλου δεν ισχύει αυτό. Γι' αυτό τώρα έχουμε τα δαχτυλικά αποτυπώματα που θα λαμβάνονται. Το Δουβλίνο προσκρούει σε αρνήσεις για ευλογές αιτίε. Τώρα η χώρες ε, από το οργανισμό του Δουβλίνου επιβαρύνονται πάρα πολύ. Τώρα, για τα δακτυλικά αποτυπώματα είδα ότι αυτά μπορεί να λαμβάνονται υποχρεωτικά. Υποχρεωτική λήψη αποτυπωμάτων δακτυλικών. Και δηλαδή θα μπορεί να είναι δυνατή άσκηση τη βίας αναφέρεται ελάχιστη, ελάχιστο επίπεδο βίας αυτό θα πρέπει να μπορεί να εφαρμόζεται ο καταναγκασμός ως σύστατο μέσο. Εδώ θέλω εξηγήσεις. Γιατί σίγουρα θα δημιουργηθούν ε, προβλήματα νομικά όταν πρόκειται για εγγύους, για ε, ανηλίκους. Εκεί πώς θα το δούμε. Επίσης, ε, θα έχουμε πρόβλημα με τις υφιστάμενες οδηγίες, αν πούμε ότι θα ασκήσουμε απειλή βία σε έναν ε, ανήλικο. Τώρα, οι 20.000 και οι 40.000. Το πρόγραμμα με την κατάσταση υπάρχει χρόνια, είναι εθελοντικό πρόγραμμα, προαιρετικό, το οποίο δεν αξιοποιείται ή δεν αξιοποιείται σχεδόν καθόλου. Δεν είναι τίποτα καινούριο δηλαδή. Και ξαφνικά τώρα μιλάμε για 40.000. Οι 60.000 ανθρώπους που πρέπει να έρθουν εδώ, να μετεγκατασταθούν, να επανεγκατασταθούν. Ε, τα κράτη-μέλη τι λένε για όλα αυτά και πώς θα πιστούν να επιδείξουν αλληλεγγύη μετά από ένα πρόγραμμα προαιρετικό. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Και επανέρχομαι στην Ελλάδα. Αν αυξάνεται ο αριθμός των προσφύγων στα νησιά τους, τι μέτρα στήριξης θα παράσχεται. Sorry, my microphone wasn't working. I Συγγνώμη, το μικρόφωνο δεν δούλευε. Λόρα Φερέρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα αδύναμα σημεία νομίζω ότι υπογραμμίστηκαν σαφώς. Γελίο είναι το νούμερο και για την Ιταλία και για την Ελλάδα. Αναφερόμαστε μόνο σε Ερυθρέα και Συρία δεν σταματάν οι, οι βάρκες. Φτάνουν εκατοντάδες βάρκες στις ακτές της Ιταλίας. αναφερόμαστε στους α, ε, μετανάστες που φτάνουν μόνο από τις 15 Απριλίου και μετά. Και επίσης δεν υπάρχει κανένα στοιχείο υποχρεωτικότητας, έτσι. Να σας θέσω λοιπόν δύο ερωτήματα. Πρώτον, ο μηχανισμός ε, μετεγκατάστασης τι προβλέπει. Ότι η Ελλάδα και η Ιταλία θα εντοπίσουν τους μετανάστες που θα μετεγκατασταθούν και θα υποδείξουν τα εθνικά σημεία που υπάρχουν σε κάθε χώρα και περιμένουν λοιπόν απάντηση από τα άλλα κράτη-μέλη για τη διαθεσιμότητά τους για να λάβουν αυτά τα άτομα για να τους μετεγκαταστήσουν τη στιγμή που κανένα κρατό μέλο δεν απαντάει ας πούμε, σε αυτέ τις αιτήσει από την Ιταλία και την Ελλάδα. Τι γίνεται με το μηχανισμό, σταματάει, θα υπάρχει ένας μηχανισμός αυτόματο αυτόματος ή λίγη διαλύεται αυτός ο μηχανισμός. Δεν υπάρχει με την κατάσταση. Και επίσης κάτι άλλο. Γιατί δεν προσφύγαμε στην οδηγία για το temporary protection, προσωρινή προστασία. Και θεωρήσατε ότι το άρθρο 78.3 είναι νομική βάση. Αν συγκρίνουμε τις, προ... τις ε, διαδικασίες είναι πολύ παρόμοιες. Αλλά στο temporary protection ε, είναι κάτι... υπάρχει κάτι το οποίο μου... μου κάνει εντύπωση. Δεν εφαρμόστηκε ποτέ μέχρι στιγμής. Είναι υποχρεωτική όμως αυτή η προσωρινή προστασία για όλα τα κράτη-μέλη και θα μας έχει επιτρέψει να ξεπεράσουμε αυτό το αδιέξοδο στο οποίο βρισκόμαστε τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δύο μέρα. Gracias, señor Τηλεγραφικά, Πρόεδρε. Από τις 8 προτεραιότητες που υπάρχουν στο θεματολόγιο, μόνο η πρώτη, ε, το να σώσουμε ζωές, είναι νομικά δεσμευτικό με βάση το 78-3. Ε, κατεπίγουσα δηλαδή περίπτωση. Το να σώσουμε ζωές. Κύριε Ρόουτε, η Euromed είναι η μόνη στρατιωτική δύναμη Ποιο ε, Ποιος λειτουργεί, ε, διάφορε ε, ΜΚΟ, οι γιατροί χωρί σύνορα. Υπάρχουν μόνο έξι εμπειρογνώμονε επίσης από έξι χώρε. Ποιο συντονίζει. Δεύτερη ερώτηση. Σήμερα το πρωί ένα νέο. Η αγαπημένη μου Μισελ Κόνιξ είπε ότι στο Europress ότι η Eurojust επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν ε, μέλη του ISIS, του Ισλαμικού κράτου, ε, κράτους, που μπαίνουν στην Ευρώπη μέσω ε, της ε, παράνομης μετανάστευσης. Πο, πολλά άτομα. άτομα έχουν ε, διεισδύσει στην Ευρώπη. Διεισδύουν με διάφορους τρόπους. Η ατζέντα προβλέπει τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ που τηρείτε το χρόνο σας. Η κυρία Μέιερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα αριθμητικά στοιχεία είναι τρομακτικά. 37.000 ε, παράνομοι μετανάστες έφτασαν στις χώρες μας τους δύο τελευταίους μήνες μέσω της Μεσογείου. Θα πρέπει να τους βοηθήσουμε περισσότερο. Διασώσαμε πολλές ζωές, πολύ καλό αυτό, αλλά θα έπρεπε να έχουμε διασώσει ακόμα περισσότερους. Και αυτό το καθήκον δεν βαραίνει τις ιδιωτικές εταιρείες, εμείς πρέπει να το κάνουμε. Η Αυστρία αρνείται πλέον να επεξεργαστεί αιτήσει ασύλου και άλλες χώρες κλείνουν τα σύνορά τους. Θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε δραστικά. Ας κοιτάξουμε το αυστραλιανό μοντέλο πολύ προσεκτικά. Το άλλο, το θέμα των προτιμήσεων των μεταναστών. Πώς πιστεύετε ότι θα λειτουργήσει κάτι τέτοιο. Δεν πιστεύετε ότι θα έχουν όλες τις ίδιες προτιμήσεις. Σουηδία, Ολλανδία και Γερμανία για παράδειγμα. Ευχαριστώ κύριο Τιπρέ. Πρόεδρε, τηλεγραφικά. Πρώτον, κείμενο του άρθρου 5, κριτήρια επιλογής μιλούμε ότι θα γίνουν μεταφορές ε, στοιχείων από ε, μια χώρα σε μια άλλη ε, και ότι θα μεταφέρουμε και ανθρώπους θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι προτιμήσεις τους λοιπόν δεν είναι πράγματα οι άνθρωποι δεύτερον σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση 10.000 ευρώ για ε, επανεγκατάσταση και 6.000 για μετεγκατάσταση γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά ποια είναι η νομική βάση και ποιος ο λόγος πίσω από αυτή τη διαφορά τρίτον άρθρο 3.2 75%. Ε, ε, ποιοι είναι αυτοί. Ποιο είναι αυτό το 75%, ποιους, ποιους αφορά ακριβώς. Τέλος, μιλάμε πολύ για την Ιταλία και την Ελλάδα, αλλά κοιτάω τα νούμερα και βλέπω ότι η Ουγγαρία ε, δέχεται περίπου παρόμοιους αριθμούς. Γιατί δεν μιλούμε για την Ουγγαρία. 55.000 έχουν φτάσει εκεί τι θα γίνει με, τι θα γίνουμε με 55.000 γιατί το, αυτό το, πρόγραμμα, ε, το έκτακτο πρόγραμμα δεν την καλύπτει. Ευχαριστώ. but it's That's what counts. Thank you, Η ποιότητα μετράει. Ευχαριστώ, Jared. Η Άννα Γκόμες. Απογοήτευση από το τελευταίο συμβούλιο. Εφημισμός όμως είναι αυτό. Όσο περισσότερο ακούμε και για τα αποτελέσματα, αλλά και για τι ε, συζητήσει που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, ντρεπόμαστε. Το ερώτημα μου είναι για τι νόμιμε οδού. Εσεί είπατε, κυρία μου, ότι είναι η άλλη όψη νομίσματο αυτή για μια ε, αποτελεσματική καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης, της σωματεμπορίας κτλ. Γιατί δεν προχωρούμε, δεν υπάρχει πολιτική θέληση στα κράτη-μέλη ή υπάρχουν πρακτικά προβλήματα. Και έπειτα, υποστηρίζω απόλυτα αυτά που είπε η Σκα και τα συμπεράσματά της και τι συστάσει της. Φυσικά, ο δεσμευτικός χαρακτήρας των μηχανισμών κατάσταση και γενικά κατανομής είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι το κρίσιμο στοιχείο. Και γιατί η Κομισιόν δεν πιέζει τα κράτη-μέλη και γιατί δεν ε, εξετάζει τους ε, μηχανισμούς ε, θεώρησης ε, όπου τα κράτη-μέλη με ύποπτους τρόπους δίνουν αυτές τις χρυσές θεωρήσεις σε πλούσιους μετανάστες ενώ αποστρέφουν το βλέμμα από τους στοχούς το οποίο τους αγνοούν, το οποίο είναι και αντιευρωπαϊκό και είναι κατά της αξιοπρέπειας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εδώ μιλάμε για προγράμματα μετεγκατάστασης και διάφορους ε, μηχανισμούς επανεγκατάστασης. 40.000, 20.000 ε, για επανεγκατάσταση. Και γίνονται οι εκατοντάδες χιλιάδες των άλλων που μπαίνουν παράνομα. Δεν το έχω καταλάβει αυτό, πώς έχει κατάσταση. Αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε είναι να θεσπίσουμε πολιτικές. Στη χώρα μου στη Σουηδία δεχόμαστε μετανάστες από τη Συρία συνεχώς και από άλλες χώρες. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν να κάνουμε είναι να δούμε ποιοι έρχονται, να τους αναγνωρίσουμε. Ξέρουμε ότι έρχονται αυτοί οι άνθρωποι κατανέμονται σε όλη την ε, Ευρώπη αλλά οι τζιχαντιστές ε, δεν είναι βέβαια ε, άνθρωποι που θέλουμε να τους έχουμε πώς θα τους ταυτοποιούμε Ίσως θα έπρεπε δηλαδή σε ορισμένε περιπτώσεις να γυρίζουν πίσω να επιστρέφουν αυτοί οι άνθρωποι Μπάρμπαρα Σπινέλη Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η απογοήτευσή μου είναι απίστευτη και για, τα νούμερα, αλλά, δηλαδή το ποσοτικό στοιχείο, αλλά και το ποιοτικό. Καταρχάς, το ποσοτικό στοιχείο. Στην Ιταλία το 2014 φτάσανε 170.000 μετανάστες και αιτούντες άσυλο. Και η μετεγκατάσταση 24.000 ανθρώπων είναι γελίο νούμερο είναι ένα σύστημα το οποίο δεν λειτουργεί ούτε για την Ιταλία, ούτε για την Ελλάδα, ούτε για την Ουγγαρία. Συμφωνώ με αυτά που υπόθηκαν σχετικά με την Ουγγαρία. Τι σκοπεύουν να κάνουν τα κρατημέλη, θα ήθελα να ξέρω. Και τι θα κάνει το Συμβούλιο μαζί με τα Συμβούλια. Και αν τα, τα, τα κράτη-μέλη ε, αρνηθούν ε, τις τα δεσμευτικά μέτρα, τι θα γίνει, χωρίς να... τι μπορούμε να κάνουμε χωρίς να αλλάξουμε το, το σύστημα του Δουβλίνου. Επίση, συμφωνώ με τη Σκά Κέλλερ ότι θα πρέπει να δοθεί βασική προτεραιότητα στι προτιμήσει των ετούντων άσυλο. Να σκεφτούμε, α πούμε, και την διευρυμένη επανένωση μια οικογένεια. ή μάλλον την επανένωση μια διευρυμένη οικογένεια. Αυτόν τον τρόπο θα αποφύγουμε και τι λεγόμενε δευτερογενεί μετακινήσεις. Ίσως και αυτό θα πρέπει να το δούμε στα πλαίσια μιας ανθεώρησης του συστήματος του Δουβλίνου. Κάτι την άποψή μου. Ευχαριστώ. Και εμείς ε, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε συνάδελφοι που ήσασταν πολύ α, σύντομοι και τα λέτε και πολύ καλά. Ηλιάνα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαι σκιώδη συγγήτρια στην έκθεση τη κυρία Κέλλερ. Το σχέδιο με την κατάσταση της Κομισιόν για την Ιταλία και την Ελλάδα Καταρχά, συνάδελφοι, α σκεφτούμε, κατα... ας μην λάβουμε υπόψη μα την ποσόστοση. Ας μιλήσουμε για την κλίδα κατανομής. Οι ποσοστώσει δεν έχουν νόημα όταν μιλάμε για ανθρώπους και κυρίως θύματα πολέμων και σειράξεων. Συμφωνώ με άλλους ότι θα πρέπει να υπάρχει το υποχρεωτικό στοιχείο. Και κύριε Ρόιτε, μην υποχωρήσετε, μην υπαναχωρήσετε από την, ε, τον υποχρεωτικό χαρακτήρα των μέτρων. Οτιδήποτε είναι θελοντικό δεν λειτουργεί και αυτό το έχουμε δει στην πράξη. Επίσης συμφωνώ ότι αυτή η κλίδα κατανομής θα πρέπει να υπακούει τον τύπο της Κομισιόν. Αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε και μόνιμες ε, λύσεις στο μέλλον. Γιατί να μην λάβουμε, ας πούμε, στον τύπο αυτό και το, την έκταση της χώρας καθώς και τον αριθμό των μεταναστών που έχουν ήδη γίνει δεκτοί στη χώρα αυτή. Επίσης, να σας ρωτήσω, έχει ξεκάθαρη άποψη η Κομισιόν για τους, χρή... για τους... Για τις, ε, τους όρους που χρησιμοποιεί μερικές φορές. Τι θα πει μαζική ας πούμε εισρωή, ε, έντονη μεταναστευτική πίεση, εθνίδια ε, εισρωή. Όλα αυτά αφορούν το άρθρο 78 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά αυτή η μαζική εισρωή είναι ένα πράγμα στην Ιταλία και τελείω διαφορετικό σε μια μικρή χώρα όπως η Βουλγαρία. Και μια άλλη δυσκολία προκύπτει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει μια σαφή διευθέτηση για τη μετεγκατάσταση των ετούντων άσυλων. Συμφωνώ με την ιδέα που ακούστηκε από τους συναδέλφους ότι οι μετανάστες θα πρέπει να δώσουν την άποψή τους, να πούν ποιες είναι οι προτιμήσεις τους, να ληφθεί υπόψη το στοιχείο της οικογενειακής, ε, οικογενειακής επανένωσης, ε, το θέμα της γλώσσας κτλ. Αλλά μην ξεχνάμε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να στρέψουμε την ισορροπία κατανομής με λάθος τρόπος. κάτι ε, κράτη-μέλη που αποκλείεται να είναι θελοντές ας πούμε για να δεχτούν μετανάστες και μετανάστες αποκλείεται να δεχτούν να πάνε εκεί. Όλα αυτά που λέτε είναι όλα πολύ χρονοβόρα, πολύ ε, δύσκολα. Και μια άλλη βασική ερώτηση. Υπάρχει μια αντίστροφη επίπτωση αυτών που προτείνεται. Αν κάποιος έχει μετεγκατασταθεί ας πούμε και αποφασίσει ότι θέλει να επιστρέψει στην χώρα προέλευσής του όταν εξομαλυθούν τα πράγματα. Και τι, τι θα γίνει γι' αυτό και επιπλέον να μου πείτε και δύο λόγια για τις, να, τις θεωρήσεις. Κάποιος άλλος. Είσαστε σκιώδης εισηγητής, γι' αυτό σας έδωσα έξτρα χρόνο. Αλλά σας παρακαλώ οι υπόλοιποι να σεβαστείτε το χρονοδιάγραμμα. Η Helga Stevens. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, μερικά σύντομα σχόλια. Να ευχαριστήσω την εισηγητρία για αυτή την ενδιαφέρουσα έκθεση. Αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν να ληφθούν υπόψη οι προτιμήσεις των ετούντων άσυλων στην πράξη. Πώς θα λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Πώς θα αποφύγουμε όλοι οι ετούντες άσυλο να διαλέγουν τις ίδιες δημοφιλείς χώρες ε, και να αφήνουν στην άκρη τις υπόλοιπες. Αυτό δεν θα αποτελούσε πραγματική αλληλεγγύη. Ασφαλώς να λάβουμε υπόψη τις ε, προτιμήσεις, αλλά έχω την εντύπωση ότι στην πράξη ίσως δεν είναι κατορθωτό. Πώς θα λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Αν πρόκειται να λάβουμε υπόψη τις προτιμήσεις, τότε ε, απομακρυνόμαστε από την Σύμβαση Γενέβης, διότι αυτή αναφέρει πως όσοι φεύγουν από περιοχές βίας ή πολέμου θα πρέπει να προστατεύονται. Αυτό είναι το σημαντικό και αυτό πρέπει να γίνει. Ε, με αυτόν τον τρόπο χάνεται λίγο η αρχική ιδέα. Πιστεύω ότι το σύστημα θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικής εφαρμογής, δεσμευτικό, είναι ο μόνος τρόπος να ε, κατανέμονται δίκαια τα βάρη. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη πόσοι, πόσοι σε άσυλο ε, βρίσκονται σε, κάποια, σε οποιαδήποτε χώρα εκείνη τη στιγμή, πόσο γιατί έχουν γίνει δεκτές στο παρελθόν κλπ. Και μια ερώτηση για το σύστημα του Δουβλίνου. Συνήθως ε, όταν σε ετών άσυλο φτάνει κάπου, καταγράφεται ε, και παρακολουθείτε. Όμως, όταν ε, πανεγκατασταθεί μετά είναι δύσκολο να επιστραφεί στην πρώτη χώρα στην οποία έφτασε. Ε, για παράδειγμα στην Ελλάδα. Θα είναι δυνατή μια τέτοια επιστροφή στη χώρα άφηξης όταν έχει πανεγκατασταθεί κάποιος. Ευχαριστώ. Ελισλάιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπε η συγγήτρια και την ευχαριστώ για τη θαυμάσια δουλειά που έκανε. Διάβασα ότι το αποτέλεσμα του Συμβουλίου ήταν απόλυτα απογοητευτικό. Πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα, λαμβάνοντα υπόψη τα... το διακύβευμα των ροών. Αν η Ευρώπη μπορεί να αντιμετωπίσει 26.000 που έλαβε χθε. Δεν ξεχνάτε ότι ο Λίβανος ε, πήρε από τη, ε, από τη Συρία ένα εκατομμύριο πρόσφυγες. Επίσης, ε, τα κράτη-μέλη μόνο το 7% όλων των νούμερων δέχονται. Αυτή είναι η αλληλεγγύη του άρθρου 78. Εδώ ζητάμε απλώς να εφαρμόσουμε τις συνθήκες μας δεν τις εφαρμόζουμε. Εφόσον τις εφαρμόζουμε, τις παραβιάζουμε. Ή το ένα ή το άλλο. Φυσικά, περιμένουμε την Κομισιόν να κάνει αυτές τις προτάσεις, να καταστήσει αυτόν το μηχανισμό μόνιμο στο μέλλον. Είναι σημαντικό να εστιάσουμε στο να λάβουμε υπόψη τις ε, προτιμήσεις των ετών των άσυλων, ιδίως όταν έχουν ε, οικογένειες και δικτύωση σε κάποια κρατημέλη που μπορούν να τους βοηθήσουν όταν φτάσουν. Δεν θα ήταν αποδεκτό να βάλουμε ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν από φυλακές σε μια άλλη φυλακή. Δεν θα πρέπει να πληρώσουν αυτοί για την έλλειψη εμπιστοσύνη που έχουν ε, τα κράτη-μέλη μεταξύ του. Κράτη-μέλη που, by the way, ε, ανήκουν στην ίδια ένωση. Παρακαλώ, 1,5 λεπτό σα παρακαλώ, συναδελφοί. Όχι παραπάνω από 1,5 λεπτό ο καθένα. Ο κύριος Λεμπρετών. Λεμπρετών, συγγνώμη. Τα ευρωπαϊκά κράτη είναι ευαίσθητα έναντι των πνιγμένων στη Μεσόγειο μεταναστών, αλλά ανησυχούν επίσης και για τις μεγάλες ροές. Ε, ένα εκατομμύριο, τουλάχιστον ένα εκατομμύριο άτομα περιμένουν στη Λιβύη για να διασχίσουν τη Μεσόγειο. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση δεν αρκεί να μιλάμε για την ανθρωπιστική πτυχή για την οποία μιλήσαμε αρκετά σήμερα. Θα πρέπει να προβλέψουμε και ένα αποτρεπτικό στοιχείο στην ευρωπαϊκή πολιτική ε, μέσω της καταπολέμησης των δικτύων διακινητών, ε, τα οποία αναφέρθηκαν αλλά μόνο κροθυγός. Ε, θα πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε τους πληθυσμούς, τον πληθυσμό σε ό,τι αφορά αυτά τα δίκτυα. Ε, αυτό ελέγχθη, αλλά δεν αρκεί. Θα πρέπει να διαπραγματευτούμε την Τουρκία, για παράδειγμα, έτσι ώστε να μην επιτρέπει να περνούν πλοία προ την κατεύθυνσή μα. Η Τουρκία είναι μεγάλη χώρα, μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση και αυτά τα δίκτυα. Επίση, θα πρέπει να δούμε αν μπορούμε να καταστρέψουμε τα ε, σκάφη των διακινητών στη Λιβύη και αν χρειαστεί να περάσουμε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, αν απαραίτητο. Δεν μιλώ για κάτι ακόμα πιο ακραίο, όπως για παράδειγμα να επιστρέφουμε κάποιους μετανάστες όπως κάνει η Αυστραλία. Η ανθρωπιστική πτυχή ασφαλώς θα πρέπει να λυθεί υπόψη βέβαια. Μιλήσαμε για επανεγκατάσταση 40.000 ατόμων που έφτασαν φέτος και μετά 20.000 κάθε χρόνο. Όλα αυτά είναι λίγα βέβαια, ως νούμερα είναι μικρά. Ε, ε, λέει η κυρία Κέλλερ. Ε, εγώ δεν θέλω να επαναγκαταστήσουμε περισσότερους, αλλά θέλω να ε, καταγγείλω ότι δίνεται λάθος στοιχεία στην κοινή γνώμη. Τα πραγματικά αθνητικά στοιχεία τα ανακοίνωσε ο Επίτροπος Αβραμόπουλος. Είπε ότι ε, μας λείπουν 50 εκατομμύρια άτομα από τον πληθυσμό μας, οπότε η μετανάστευση μπορεί να είναι μια λύση. Οπότε πόσα είναι τελικά τα πραγματικά, ε, οι πραγματικές μας ανάγκες, τα πραγματικά νούμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, θα είμαι σύντομη. Συμφωνώ με αυτούς που λένε ότι είναι τρομερό που δεν είναι δεσμευτικός ο μηχανισμός μετά από συμφωνία. Η ε, αλληλεγγύη δεν περιορίζεται μόνο στα διαφορετικά ταμεία, πρέπει να επεκτείνεται και στη διάσωση ζώων. Ελπίζω ότι στο πρόγραμμα αυτό της μετεγκατάστασης που προτείνεται θα έρθουν και άλλα κράτη-μέλη, αλλά δεν αρκεί όμως είναι για 40.000 ανθρώπους, δεν αρκεί. Θέλω επίσης να πω ότι είναι μια εποχή τώρα στην Ευρώπη που χρειαζόμαστε ηγεσία, πολιτικούς, βουλευτές, πρωθυπουργούς, όχι λαϊκιστές, αλλά ανθρώπους που καταλαβαίνουν και εξηγούν ότι χρειαζόμαστε χέρια εργατικά, θέλουμε ε, να αλλάξουμε τα δημογραφικά μας δεδομένα. Θέλουμε πολλούς ξένους, θέλουμε ειδικευμένου, γιατί έτσι μπορεί να αλλάξει ε, το ευρωπαϊκό αφήγημα. Πολλοί αντιμετωπίζονται άσχημα, πολλοί δαιμονοποιούνται γιατί έρχονται από εμπόλεμες περιοχές. Ντρέπομαι γι' αυτό. Να σας ρωτήσω και κάτι για τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Υπάρχει απόφαση του δικαστηρίου και το ε, Κοινοβούλιο ήταν σαφές σε σχέση με το κανονισμό του Δουβλίνου. Το Συμβούλιο όμως διαφοροποιείται με τρόπο απαράδεκτο, γιατί εδώ πρόκειται για ασυνόδευτους ανηλίκους. Δεν μπορεί να τους πηγαίνω φέρνουμε και να τους θέλουμε τόθη κήθε στα κράτη-μέλη. Εσάς η πρότασή σας πώς επηρεάζει την αντιμετώπιση των ασυνόδευτων ανηλίκων. Ευχαριστώ. Κάποιοι συνάδελφοι ε, έδωσαν αργότερα μήνυμα ότι θέλουν να λάβουν το λόγο. Ε, είναι δύσκολο αυτό. Λοιπόν, έχουμε δύο ακόμα μιλητές. Ε, θα, θα να φεύγουν μετά. Ίσως ένα δεύτερο γύρο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ που αποσύρεστε. Για να ακούσουμε τώρα το Γενικό Διευθυντή. Τι θα μας απαντήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 20 ερωτήσει άκουσα. Εάν πρέπει να απαντήσω και στι 20, θα χρειαζόμουν το διπλάσιο χρόνο. Γι' αυτό θα είμαι λακωνικός και θα πω. Πρώτον, χρειαζόμαστε ένα νομικά δεσμευτικό κείμενο, μια νομικά δεσμευτική πρόταση για να λειτουργήσει το πράγμα και το κατάλαβαν τα κράτη-μέλη. Εδώ μιλάμε για τη λίγα κατανομής, τα νούμερα, αλλά δεν μιλάμε για την ε, νομικά δεσμευτική πρόταση η οποία θεσπίζει το σύστημα, καθορίζει την αλληλεπίδραση μεταξύ των κρατών μελών και πώς λαμβάνει η χώρα ή μιλάει για τις προτιμήσεις και πώς μπορούν να ενσωματωθούν στο σύστημα για να αποφύγουμε και τις δευτερογενείς μετακινήσεις. Μια προληπτική ας πούμε, στάση στις ε, δευτερογενείς μετακινήσεις παρά μια κατασταλτική προσέγγιση. Και ελπίζω λοιπόν και στις συζητήσεις στο Συμβούλιο να βρούμε και κάποια κοινά σημεία επ' αυτού. Συμφωνώ με όλους σας ότι τα νούμερα είναι πάρα πολύ μικρά σε σχέση με την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε. Παράλληλα όμως, σας καλώ να σκεφτείτε ότι στην πράξη πρώτη φορά κάνουμε κάτι τέτοιο. Έτσι. Ποτέ δεν έχουμε ξανακάνει τέτοια πρόταση. Είναι μια πρωτιά αυτή. Και γι' αυτό είμαι και περήφανος που δουλεύω στην Κομισιόν ε, υπό ένα πρόεδρο, υπό έναν ηγέτη Κομισιόν που δείχνει τέτοιο, τέτοια ηγετική ικανότητα. Επίσης, ο κύριο Ντεπχέ έκανε μια συγκεκριμένη ερώτηση, το 75% αυτό το περίφημο, ε, για τους Ερυθρέους και για τους Σύριους. 6.000, 10.000. για το Ταμείο Ασύλου οι 10.000 ε, ενσωματωμένοι, ενώ το, το 6.000 δεν καλύπτει τα, δηλαδή καλύπτει και τα έξοδα μεταφοράς, τα 6.000 είναι χωρί τα έξοδα μεταφοράς. Το θέμα των ανησυχιών περί ασφάλειας. Αυτό ε, λαμβάνεται υπόψη στην απόφαση. Ε, δημόσια τάξη, δημόσια ασφάλεια. Είναι λόγοι άρνησης για τα κράτη-μέλη. Και δημιουργούμε ένα σύστημα ε, όπου υπάρχει έλεγχος, υπάρχει, υπάρχουν αυτά και τα hot spot και στα πλαίσια του μηχανισμού μετεγκατάστασης η Frontex θα εμπλακεί, η Europol, ούτω ώστε να λάβουμε υπόψη μας όλα τα θέματα ασφαλείας. Εάν κοιτούσαμε απλώς τις προτιμήσεις, θα είμαστε σε επίπεδο γιουρίμα της Μάλτας. Αλλά δεν γίνεται να το κάνουμε αυτό. Θα πάρουμε υπόψη, θα λάβουμε υπόψη όσο μπορούμε τις ε, προτιμήσεις, όχι παραπάνω. Ασυνόδευτη ανήλικη, τελευταίο θέμα. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο της απόφασης και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο γι' αυτό και ελπίζω στο δεύτερο εξάμεινο του 2015 με τη βοήθεια της Λουξεμβουργιάζικης Προεδρίας θα βρούμε λύσεις για το θέμα των συνόδευτων ανηλίκων στα πλαίσια του κανονισμού του Δουβλίνου. Νομικά στοιχεία, νομικές αποδείξεις. Η επανεγκατάσταση είναι μία νόμιμη οδός. Δίνουμε 20.000 θέσεις σε ανθρώπους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να έρθουν στην Ευρώπη, να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία βασική προσέγγιση. Δεύτερη, στο συνολικό πλαίσιο της νόμιμης μετανάστευσης, δεν θα μπω τώρα βέβαια σε λεπτομέρειες ερευνητών, μπλε κάρτας, εποχιακών ε, εργαζομένων, τι θα κάνουμε του χρόνου, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε. Εγώ αυτό που προσπάθησα να σας πω είναι ότι η Ευρώπη θα πρέπει να είναι σημείο αναφοράς σε ό,τι αφορά την νόμιμη μετανάστευση. Μίλησαμε για το καναδικό και όπως το καναδικό σύστημα είναι έτσι πρότυπο ας πούμε, έτσι θα θέλω, να είναι και το ευρωπαϊκό σύστημα. Ε, αλλά θα ήθελα να κάνω αυτή τη συζήτηση για την νόμιμη μετανάστευση έτσι πιο ενδελεχώς μαζί σας. Τα hot spots τα κάλυψα. Σας παρακαλώ. Υπάρχουν πάρα πολλά σχόλια, πάρα πολλές συνεισφορές. Εδώ μοιραζόμαστε το μικρόφωνο εδώ με τον τη Κομισιόν. Υπάρχουν τόσε πολλέ ε, ερωτήσει. έχει κατακλειστεί ο, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Έτσι αντιμετωπίζουμε εμεί του επιτρόπου, έτσι. Ε, σας παρακαλώ, συνάδελφοι, μόνο αν έχετε ε, έξτρα σημεία πολύ συγκεκριμένα που δεν έχουν ακουστεί, μόνο τότε θα σα δώσω, γιατί έχουμε πολύ λίγα λεφτά ακόμα. Δεν απαντήσετε στο ερώτημά μου για την Ουγγαρία. Γιατί? Γιατί και όχι, όχι και η Ουγγαρία. Τι θα κάνουμε με την Ουγγαρία. Ε, καταρχήν σας πω ότι συζητήσαμε με την Ουγγαρία και όταν υποβάλαμε την πρόταση η κατάσταση στην Ουγγαρία ήταν διαφορετική. Δεύτερον, αν δείτε τα νούμερα, στην Ουγγαρία έχουμε 27 περίπου χιλιάδες ε, που προστίθενται οι οποίοι θα πρέπει να επιστρέψουν Παρακολουθώ όμω πολύ στενά την κατάσταση στην Ουγγαρία και η πρόταση απόφασης μάλλον και θα ληφθεί μια καινούργια απόφαση για την Ουγγαρία ειδικά αν η κατάσταση επιδεινωθεί. Ευχαριστώ. Μ' αρέσει αυτό το ανακριτικό ύφος. Μην ανησυχείτε, Πρόεδρε. Ε, Κορνίλια σε αντίθεση με άλλους, εγώ είχα ρωτήσει για τα αποτυπώματα που υπάρχουν νομικές επιφυλάξεις, αν όχι από εμάς, ίσως από άλλους. Κοιτάξτε, στις κατευθυντήριες γραμμές μας προσπαθήσαμε να λάβουμε υπόψη μας και να περιγράψουμε την πρακτική στα κράτη-μέλη. Αυτή που αναφέρατε είναι η πρακτική κράτους μέλους γνωστού στη Σουηδία, που επιτρέπει σε ορισμένες συνθήκες και ε, ε, ε, λαμβάνοντας και αναλογικά να λαμβάνονται βιαίως τα αποτυπώματα γιατί τα δακτυλικά αποτυπώματα πρέπει να υπάρχουν και αν κάποιος αρνηθεί τη λήψη των αποτυπωμάτων αυτών πρέπει να προβλεφθούν στις κατευθυντήριες γραμμές διάφορες μέθοδοι για να ληφθούν. Ναι, ίσως δεν σας ε, καλύπτει αυτό. Εγώ ε, τώρα δεν σας ζητώ να κάνετε και άλλες ερωτήσεις, μόνο διευκρινιστικές. Ορίστε. Κυρία Κίνγκε. Δεν άκουσα την απάντηση στο ερώτημα για, ε, για τον επαναπατρισμό. Είχα ρωτήσει το εξή η Κομισιόν έχει πάρει προληπτικά μέτρα για να εμποδίσει κάποια κράτη-μέλη να υλοποιήσουν πολιτικές επαναπατρισμού που μπορούν να ζημιώσουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες και δικαιώματα των ανθρώπων. Yes, of course we have... Uh, Έχουμε την οδηγία επιστροφής η οποία προβλέπει συγκεκριμένες και σαφείς διαδικασίες. και οποιοδήποτε κράτος μέλος ε, δεν την εφαρμόζει το ε, κινούμε διαδικασία παραβάση εναντίον του. Ευχαριστούμε πολύ λέει ο Πρόεδρος για αυτή την παρουσίαση και για τις απαντήσεις. Θέλω να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους για την συμμετοχή τους και για τα σχόλιά τους τόσο για την έκθεση Σκακελέρ όσο και για τις προτάσεις κομισιών. και η Προεδρία νομίζω του Λουξεμβούργου ε, θα βρει και πολύ χρήσιμη αυτή τη συζήτηση εν ώψη του Συμβουλίου, του Συμβουλίου της Πέμπτης. Ελπίζουμε ότι την Πέμπτη θα δούμε κάποιο από το αποτέλεσμα, θα είμαστε παρόντες, θα εκπροσωπήσουμε την εκπροσωπή πολύ δυναμικά με απόψεις που θα βασίζονται σε μεγάλο βαθμό και στα σημερινά σχόλια. Η σημερινή ενημέρωση ήταν πραγματικά πολύτιμη. Περνάμε στην κατάσταση της Μεσογείου. Ε, έκθεση Τσόλα και Κιέγγε. Είναι μια συγκεκριμένη περιοχή πάρα πολύ σημαντική. Τη συζητήσαμε ήδη και ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει το θέμα των πλειοκτητών. Ε, έχουμε τον Γενικό Διευθυντή της Νορβηγικής Ένωσης Πλειοκτητών μαζί μας. Ε, και άλλον έναν ε, καλεσμένο που περιμένουν. Πρόκειται για μια παρουσίαση 10 λεπτών θα, δούμε θα ακούσουμε τον κύριο Χέντριξον ή τον Πάτρικ πρώτα. Πρώτα θα μιλήσει ο Πάτρικ Φερχόβεν, ε, γενικός ε, ε, γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πλειοκτητών και μετά θα ακούσουμε τον ε, νορβηγό εκπρόσωπο των πλειοκτητών. Παρακαλώ, έχετε το λόγο και σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μοιραζόμαστε το μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ πολύ που μας καλέσατε. Εκπροσωπώ την ΕΞΑ, την Ευρωπαϊκή για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση Πλειοκτητών. Πρόκειται για μια οργάνωση ομπρέλα που εκπροσωπεί όλες τις ενώσεις, όλους τους συλλόγους ε, ε, πλειοκτητών της Ευρώπης. Ο Στούλα Έριξον είναι ο Γενικός Διευθυντής της Νορβηγικής Ένωσης Πλειοκτητών. Ε, θα με συνοδεύσει. Καταρχήν να σας μιλήσω, για θα μιλήσω εγώ καταρχήν για κάποια αριθμητικά στοιχεία και μετά ο συνάδελφός μου θα σας δείξει ένα βίντεο και θα σας μιλήσει για κάποιες ανησυχίες που έχουμε για το ρόλο μας. Ε, καταρχήν, γιατί είμαστε εδώ σήμερα ως πλειοκτήτες. Ποιος είναι ο ρόλος μας τη διάσωση των μεταναστών στη θάλασσα. Ε, μετά την κλιμάκωση της ε, κρίσης ε, στη Μεσόγειο από την αρχή του 2014, ε, εκτιμήσαμε ότι 1.200 εμπορικά σκάφη ενεπλάξαν σε, διάσω, επιχείρηση διάσωσης. Η βοήθεια των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα στη θάλασσα είναι τμήμα του ηθικού κώδικα των σκαφών αλλά και δράζεται και στο διεθνές δίκαιο. Αυτή η παράδοση όμως και αυτός ο κώδικας ε, δεν είχε ποτέ ε, σχεδιαστεί για την διάσωση τόσο μεγάλων αριθμών. Γνωρίζετε τα στατιστικά πολύ καλύτερα από ότι εμείς. Ε, οι ροές έχουν αυξηθεί πάρα πολύ από το 2013 και μέσα στο 2014. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Αυτή εδώ η διαφάνεια μας δείχνει την εμπλοκή της του εμπορικού ναυτικού. Μιλάμε για το 2014, νούμερο του 2014 που μας τα έδωσε η Ιταλική Ακτοφυλακή. Ε, το 2014 μέχρι τον Οκτώβριο του 2014 η, Ιταλία διατηρούσε την Mare Nostrum που ήταν μια ε, ευρεία επιχείρηση διάσωσης που διέσωσε το 50% περίπου ε, των μεταναστών. Παρ' όλα αυτά πάνω από 35% ήταν η δική μας συνεισφορά, δηλαδή διασώσαμε πάνω από 35% των μεταναστών με εμπορικά σκάφη. Επόμενη διαφάνεια, αυτή είναι η κατάσταση σήμερα, φέτος μάλλον, μέχρι τις 10 Ιουνίου. Βλέπετε ότι ο εμπορικός στόλος ε, αύξησε τη συμμετοχή του. Ε, γύρω στο Πάσχα ε, χτύπησαν καμπανάκια κινδύνου γιατί αυτή η κατάσταση δεν είναι βιώσιμη για το εμπορικό ναυτικό. Και όταν στα μέσα Απριλίου ε, είχαμε αυτά τα δυσάρεστα επεισόδια, ε, το Συμβούλιο Τριπλασίας τον προπολογισμό των επιχειρήσεων και τη γεωγραφική κάλυψη. Το, το αποτέλεσμα αυτών το μέτρων δεν το βλέπουμε στα αριθμητικά στοιχεία γιατί η επιχείρηση τρίτον άρχισε να εφαρμόζεται από το τέλος Μαΐου και μετά. Ελπίζουμε ότι θα βοηθήσει, ε, ότι θα ανακουφίσει ε, το εμπορικό ναυτικό από το βάρος του. Τελευταία διαφάνεια, σε απόλυτα νούμερα, βλέπετε το 2014 883 πλοία κινητοποιήθηκαν για να διασώσουν μετανάστες ε, και 254 το 2015 και βλέπετε και τα άτομα τα οποία διασωσάν. Τώρα θα δώσω το λόγο στον συνάδελφό μου τον Στούρλα για να μας μιλήσει για το πρακτικό αντίκτυπο που έχει αυτή η κατάσταση στις ε, εταιρείε μας. Αλλάζουμε θέση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ε, βουλευτές, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση να παρουσιάσω τις απόψεις μας για αυτήν την κλιμακούμενη ανθρωπιστική κατάσταση. Ευχαριστώ επίσης την Επιτροπή για την ε, σημαντική πρωτοβουλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία διαθέτει πόρους ε, περισσότερους ε, για κάποιες επιχειρήσεις διάσωσης στη Μεσόγειο. Η Νορβηγία από τον Ιούνιο συμμετέχει με ένα σκάφος. Θα ήθελα να σας ε, πω δύο λόγια για τις επιχειρήσεις ε, διάσωσης Το πλοίο το περασμένο καλοκαίρι ε, εξυπηρέτησε ως πλατφόρμα το σκάφος αυτό και διέσωσε ένα πλοίο 2.000 ανθρώπους στα πλαίσια 16 διαφορετικών επιχειρήσεων διάσωσης. Κοιτάξτε εδώ αυτό το φίλμα. This is what it Αυτή είναι η εικόνα σε μια επιχείρηση διάσωσης. Νομίζω ότι το μήνυμα από αυτό το φιλμ είναι ότι ε, δεν πρόκειται για μεγάλο αριθμό διάσωσης ε, μεταναστών, προσφύγων από εμπορικά πλοία. Το πιο σημαντικό μήνυμα είναι ότι αυτές οι καταστάσεις αφορούν ανθρώπους σε κίνδυνο που διασώζονται από άλλους ανθρώπους. Είχαμε από τη Λιβύη, μία έγκυο από την Σομαλία ε, που διασωθήκε άλλους από το Μαλί. Παρακολουθούμε από κοντά τις καταστάσεις αυτές και συμμετέχουμε ενεργά. Είμαστε από τους πιο δραστήριους ε, στόλους και τώρα πάνω από 1.800 πλοία μας ε, συμμετέχουν σε όλο τον κόσμο σε επιχειρήσεις και στα ύδατα μεταξύ Ιταλίας, Μάλτας, Λιβύης, ε, Συρίας. Και αυτά ε, είναι επιχειρήσεις ε, διάσωσης που πολλές φορές συνδυάζονται και με κατάπλουσε λιμάνια της περιοχής. Το 2014 τα εμπορικά σκάφη διέσωσαν πάνω από 40.000 μετανάστες, δηλαδή έναν στους πέντε του συνόλου των ανθρώπων που διασώθησαν στην Μεσόγειο και το 2015 παρόμοια είναι τα στοιχεία και δείχνουν ότι ο συνολικός αριθμός των μεταναστών αυξάνεται κάθετα. Να είμαι απόλυτα σαφής και να πω ότι οι εταιρείε μέλη και οι NSA θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις αυτές Είμαστε περήφανοι για την παράδοσή μας στο εμπορικό ναυτικό και είναι και νομική μας ευθύνη, ευθύνη που απορρέει από το δίκαιο. Η αντιμετώπιση αυτής της ανθρωπιστικής καταστροφής μεγάλης κλίμακας ε, θα πρέπει να βρίσκεται στα χέρια της διεθνούς κοινότητας ε, και στα κυρίαρχα κράτη. Για πολύ καιρό η Ευρώπη είχε στρέψει την ε, πλάτη στην Μεσόγειο και μόνο στο εμπορικό στόλο και η Ιταλία αντιμετώπιζαν το πρόβλημα. Πρέπει εδώ να εκφράσουμε το σεβασμό μας και την εκτίμησή μας για τι τις δυνατότητες που προσφέρθηκαν και την αποτελεσματικότητα του Ιταλικού ναυτικού και ακτοφυλακή λιμεναρχείων. Ε, τα πλοία μας θα συνεχίσουν να συμπαρίστανται τα εμπορικά ε, σκάφη όμως δεν μπορούν και δεν θα έπρεπε να θεωρούνται αναπόσπαστο σημαντικό και μόνιμο κομμάτι των διαθέσιμων πόρων για επιχειρήσεις διάσωσης στην ε, Μεσόγειο. Ο βασικός λόγος γι' αυτό είναι ότι τα εμπορικά πληρώματα και τα σκάφη δεν είναι εξοπλισμένα για να συμμετέχουν σε ε, τέτοιες μεγάλες κλίμακες επιχειρήσεις διάσωσης έρευνας. Και με τις καλύτερες ε, προθέσεις και παρεμβάσεις ε, μπορεί να τεθούν σε κίνδυνο οι ζωές των, των μεταναστών, ιδιαίτερα τη νύχτα. Τα εμπορικά πλοία δεν μπορεί να έχουν την ικανότητα και τα αναγκαία μέσα για να ε, καλύψουν τις ανάγκες εν πλώ ε, μεγάλου αριθμού ατόμων ε, μέχρι να αποβιβαστούν οι άνθρωποι αυτοί. Επιπροσθέτως, αυτές οι καταστάσεις ε, δημιουργούν μεγάλα προβλήματα ε, ασφάλειας, ε, προστασίας, υγείας και τα, πολλές φορές τα πληρώματά μας δεν είναι και ψυχολογικά εκπαιδευμένα για να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους ε, δύσκολες καταστάσεις. Ε, πολλές ε, φορές βλέπουν νεκρά πτώματα οικογένειες, οικογενειών ολόκληρων να επιπλέουν στο νερό και αυτό είναι τρομερά τραυματική εμπειρία. Έχω πλήρωμα 15 ανθρώπων που δέχονται 500 ανθρώπους από διάφορες εθνότητες, θρησκείες, μικρούς, μεγάλους, μωρά ε, ορισμένοι ε, ε, νοσούν βαρύτατα, άλλοι είναι σε κατάσταση σοκ γιατί είδαν να πεθαίνει στη θάλασσα κάποιος. Άλλοι μπορεί να έχουν μεταδοτικά νοσήματα και αυτό είναι μεγάλη πρόκληση για τα πληρώματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις. Ναι, τίθενται δηλαδή θέματα και πρακτικά και νομικά και εμπορικά και εμείς ε, λειτουργούμε πάνω σε αυτή τη βάση επί 24 ώρου. Ε, πρέπει λοιπόν να λάβετε υπόψη σας ότι πρέπει να προετοιμάσουμε και το πλοίο και το πλήρωμα πριν ε, συμμετάσχουμε σε τέτοια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Οι κατευθυντήριες γραμμές ε, περιλαμβάνουν και ενημέρωση ε, πριν από την επιχείρηση με το πλήρωμα, ενημέρωση, ε, ενδείξεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σχετικά με το μετατραυματικό σοκ κλπ συχνά μας ρωτούν την γνώμη μας ε, σχετικά με το πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται η ανθρωπιστική κρίση στη Μεσόγειο. Εμείς λέμε ότι η τεράστια κλίμακα και συνθετότητα αυτού του προβλήματος απαιτεί μια διεθνή απόκριση συνεπή σφαιρική και μακροπρόθεσμη. Δεν θεωρούμε ότι ε, μια ένωση όπως η δική μας να, ε, ε, ότι επιτρέπεται να εκφράζει απόψεις σε σχέση με αυτές τις πολιτικές. Όμως για πολύ καιρό εργαστήκαμε για να ενημερώσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε και τους πολιτικούς στην Νορβηγία και τους Ευρωπαίους πολιτικούς. Επίσης υποβάλαμε πέντε συστάσεις γενικότερες που θα ήθελα να τις παρουσιάσω. Η διεθνή κοινότητα πρέπει να κινητοποιήσει πόρου ούτως ώστε να αντιμετωπίσει τη ρίζα των προβλημάτων. Ε, οι άνθρωποι ε, φεύγουν από εμφύλιο, ε, καταπίεση, φτώχεια. Οι διεθνείς ε, προσπάθειες ε, βοήθειας θα πρέπει να επικεντρώνονται στη βοήθεια ε, των ανθρώπων εκεί, στα σπίτια τους, στη χώρα τους, ούτω ώστε να τους αποτρέψουν από το να, να κάνουν αυτό το επικίνδυνο ταξίδι. Τρίτον, η διεθνής κοινότητα υποχρεούται να καταπολεμήσει τους διακινητές, τους κινητούς, που, τους ε, που θέτουν σε κίνδυνο χιλιάδες ζωές, ε, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια ότι δεν είναι όλοι οι διακινητές κακοί άνθρωποι για πολλούς, ε, συμβολίζουν την ε, δυνατότητα διαφυγής. Τέταρτον, η διεθνή κοινότητα θα πρέπει να έχει δυνατότητε διαθέσιμε για επιχειρήσει έρευνα διάσωση στη θάλασσα. Αυτό σημαίνει ότι οι ευρωπαϊκέ χώρε θα πρέπει να είναι έτοιμε να αυξήσουν τι δυνατότητε που παρέχουν, το δυναμικό του, ούτω ώστε να κλιμακώσουν την χρησιμοποίηση πλοίων γιατί αυξάνεται η μετανάσταση ε, ριζικά και ο ένας ε, στους τέσσερις ή στους πέντε ακόμα διασώζεται από εμπορικά σκάφη. Αυτό δεν είναι σωστό και θα πρέπει να βελτιωθεί από τα ευρωπαϊκά κράτη ευελιξία και να επικεντρώνουν κάθε φορά τα μέσα εκεί όπου υπάρχουν οι μεταναστευτικές ροές. Καμιά φορά αυτό είναι εκτός ε, τομέα αρμοδιότητας ευθύνης του Frontex. Ε, γιατί επίσης ε, τώρα τα στοιχεία ε, εξόδου από Τουρκία προς Ελλάδα δεν αυξάνονται τόσο ραγδαία. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ταχείας αποβίβασης των μεταναστών που διασώζονται από εμπορικά πλοία και να φάρουν στα κοντινά λιμάνια. Δεν υπάρχει μία απάντηση, μία λύση για να αντιμετωπίσει τη σύγχρονη ανθρωπιστική κρίση. Αλλά η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί παρά να δράσει σύντονα και αποφασισμένα στις προσπάθειές της. Χρειάζεται λοιπόν πρωτοβουλία σφαιρική, ε, η οποία νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό προτείνεται και από τη δική σας Επιτροπή. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. ευχαριστώ και του δύο. Το, μικρό, το δικό μου μικρόφωνο δεν δουλεύει τώρα. Σα ευχαριστώ και του δύο που ήρθατε εδώ. Φυσικά έχετε κάθε δικαίωμα να είστε παρόντες ε, και να συνεισφέρετε στην ε, έκθεση ιδιαίτερη πρωτοβουλία, τη κυρία Μετσόλα και Κιέγγε, γιατί αντιμετωπίσετε μια πολύ δύσκολη κατάσταση σε μεγάλη κλίμακα. Υπάρχει το δίκαιο της θάλασσα ε, που σας θέτει σε πολύ δύσκολη θέση και πιέστηκε χρονικά. Θα είδατε τις αντιδράσεις των συναδέλφων. Όλοι που παρακολουθούν την κατάσταση στη Μεσόγειο γνωρίζουν ότι πολλά από τα μέλη σας ε, έδρασαν με αξιοθαύμαστο τρόπο και έσωσαν ζωές. Τα εκτιμούμε αυτά τα μέλη. Ειδικά ε, με την επιχείρηση Mare Και, εκεί το εμπορικό ναυτικό στα πλαίσια του Mare Nostrum ε, βοήθησε πάρα πολύ το Ιταλικό ναυτικό και έσωσε πάρα πολλά άτομα. Ε, θα υπάρξουν πολλές ερωτήσεις ε, να ξεκινήσω με τους δύο συγητές και θα σας ζητήσω όλους να είσαστε πολύ συγκεκριμένοι και να μιλήσετε για το νομικό ηθικό δίλημα που αντιμετωπίζουν οι, οι εφοπλιστές. Και ξεκινάμε με την εισηγήτρια, την κυρία Μετσόλα. Δεν θέλω να μιλήσουμε για το έγγραφο εργασία, και την αλληλεγγύη δηλαδή και τι νόμιμε οδού, που είναι το επόμενο θέμα. Αυτό είναι το επόμενο σημείο, έτσι. Γιατί σκόπευα να τα πω όλα μαζί σε μια παρέμβαση. Είχαμε τη συζήτηση για την ευρωπαϊκή μετανάστευση και σας αντικατέστησαν ε, εκεί. Σας παρακαλώ τώρα να εστιάσουμε μόνο στην, ε, στο εμπορικό ναυτικό, στο θέμα της ναυτιλίας. Ωραία, δεν μίλησα άλλη φορά σήμερα. Πρέπει να πω και δύο λόγια και για το θέμα της μετανάστευσης. Σας ευχαριστώ πάντως ε, τον κύριο Χέριξον και τον κύριο Φερχόφεν για τις παρουσιάσεις τους, γιατί από αυτά που είδαμε στις συζητήσεις και στην όλη διαδικασία προετοιμασίας της έκθεσης είναι ότι η εμπορική ναυτιλία, το εμπορικό ναυτικό ε, κάνει πράγματα που, τα, που περνάνε Και είναι σαφές ότι ο ρόλος που παίζεται, ο οποίος είναι αξιέπαινος, δεν μπορεί να είναι μια εμβαλωματική λύση για την αδράνεια των κρατών μελών. Και εδώ μπαίνουμε στο βασικό θέμα του τι κάνουμε για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τα μέτρα αλληλεγγύης αποτελεσματικά και να εξασφαλίσουμε την νόμιμη και ασφαλή πρόσβαση στα άτομα, στα τα οποία είναι επιλέξιμα προστασίας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε και τις ε, τραγωδίες εν πλώ. Και για να μπορέσουμε να βρούμε τρόπους που θα εμποδίσουν τα άτομα τα οποία δεν έχουν άλλη λύση παρά να μπουν σε ένα σκάφος και να αντιμετωπίσουν ε, το φάσμα του θανάτου. Να το εμποδίσουμε αυτά τα άτομα και να τα βοηθήσουμε πριν να εξαναγκαστούν να προσφύγουν στους, δια... διακινητές. Ε, η επανεκατάσταση συμφωνώ ότι είναι μία ε, λύση, αλλά το κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να παίξει το ρόλο του. θα πρέπει να έχουμε μια μόνιμη λύση. Θα πρέπει να δούμε εργαλείο όπως το σύστημα ανθρωπιστικών θεωρήσεων, διευκόλυνση της πρόσβασης για φοιτητές, ε, ε, επαγγελματική κατάρτιση κτλ. από ξένους δηλαδή και η οδηγία για την προσωρινή προστασία η οποία ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκε. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να μας βοηθήσουν τόσο ώστε να μην ξανακούσουμε επιχειρήματα για την ε, φοβερή αυτή εισδροή που ξαφνικά μας κατακλείζει Έχω να πω πάρα πολλά ακόμα, αλλά θα καταλήξω ε, και ελπίζω τέλο πάντων σε μια άλλη στενδρία να την έχω. Να σα πω ότι η Άσο δεν αναφέρθηκε καθόλου σήμερα ε, όσο ήμουν εδώ. Ε, παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, θα πρέπει να ενισχυθεί αν θέλουμε να παίξει βασικό ρόλο στη θάλασσα και να εφαρμόσει την νομοθεσία του Ευρωπαϊκού Ασύλου στην ειδικά σε αυτόν τον τομέα, στη θάλασσα δηλαδή. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ Ρομπέρτα που περιορίστηκε το θέμα της ναυτιλίας. Ε, τα υπόλοιπα θέματα τα συζητήσαμε νωρίτερα. Ε, ήθελα απλώς να εστιάσουμε τώρα στην α, ναυτιλία. Λοιπόν, θα ακούσατε πάρα πολλά σχόλια. Παρακαλώ σημειώσετε αυτά στα οποία θέλετε να απαντήσετε, τα βασικά σημεία στα οποία θέλετε να απαντήσετε, ούτως ώστε να σας δώσω στο τέλος το λόγο για να πείτε και εσείς δυο λόγια. Δεν χρειάζεται να απαντήσετε σε όλα. Θα ακούσετε και πολλέ παρατηρήσει ούτω ή άλλω. Η συνεισηγήτρια είναι η επόμενη, η κυρία Κιάνγκε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ εκ νέου τον Γενικό Διευθυντή της Ένωσης ε, Εφοπλιστών και για τη συνεισφορά που ακούσαμε μόλις στη συζήτησή μας. Η προσπάθειά μας αυτούς τους ε, τελευταίους μήνες ε, μας οδήγησε σε συναντήσεις ε, και με άλλες ομάδες που ασχολούνται. Υπάρχει ανεκτήμητη βοήθεια από το εμπορικό ναυτικό και οι δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα είναι πολύτιμες. Όπως είπα και στην προηγούμενη παρέμβασή μου, θέλω ξανά να πω ότι μιλάτε για αυτό το θέμα, χαίρομαι που μιλάτε για αυτό το θέμα, αυτή η δραστηριότητα Τη ε, διάσωση, τη έρευνας και διάσωση δεν μπορούμε να την αφήσουμε σε ιδιώτε. Είναι η ευθύνη των κρατών μελών να δώσουν και τα μέσα και τη χρηματοδότηση για να εξασφαλίσουμε αυτέ τι ε, επιχειρήσει και ότι διεξάγονται σωστά. Ε, τα σημεία τα οποία πρέπει να τεθούν κατά την άποψή μου και που παρουσιάστηκαν και στην έκθεση είναι το θέμα τη εκπαίδευση των ατόμων τα οποία επιβαίνουν σε αυτά τα σκάφη, τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν και τα άτομα αλλά και, τα, και οι μετανάστες που σώζονται, γιατί δεν, υπάρχουν, ε, δεν υπάρχει γνώση, ας πούμε, πάνω σε αυτά τα σκάφη, κανένα δεν ξέρει τι να κάνει. Και επίσης δεν υπάρχουν και επαρκή σπόροι Ένα άλλο σημείο είναι το θέμα του συντονισμού μεταξύ των επιχειρήσεων των ευρωπαϊκής φύσεως και των ε, προσπαθειών που κάνει το εμπορικό ναυτικό. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το δούμε περισσότερο. Τι κάνει η Ευρώπη μαζί με το, την εμπορική ναυτιλία μαζί. Ε, Κλείνοντα, θα να σα πω ότι για να καταφέρουμε να μειώσουμε τον αριθμό των ατόμων που εμπιστεύουν τη ζωή του σε αυτέ τι παράνομε, σε αυτού του ανθρώπου και σε αυτή την της οδού, οδούς ε, χρειάζεται μια τέτοια ολιστική προσέγγιση και είναι πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία μας, νομίζω. Ευχαριστώ. Ο επόμενος, η Σεσίλια Βίξτρομ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. και στους ε, δύο εκπροσώπους των εφοπλιστών θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας ε, και τον απεριόριστο σεβασμό μας για τόσα κάνετε. Λαμβάνοντα υπόψη ότι οι άνθρωποι που διασώζουν ε, τους μετανάστες αυτούς δεν είναι εκπαιδευμένοι να κάνουν κάτι τέτοιο ούτε και έχουν παρόμοια εμπειρία. Ε, υποφέρουν από ψυχολογικά τραύματα Παρόλα αυτά, το παράδειγμα τους ε, είναι μοναδικό και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να το δουν και ιδιαίτερα τα κράτη-μέλη τα οποία αρνούνται να, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να παράσχουν ε, πόρους, πλοία και να ανοίξουν τα σύνορά τους ε, προκειμένου να δεχθούν αυτούς τους μετανάστες που χρειάζονται και έχουν δικαίωμα την διεθνούς προστασίας και μετεγκατάστασης. Πολλά θα μπορούσα να πω, αλλά εκ μέρου ε, πολλών που ήδη εγκατέλειψαν την αίθουσα χρειάστηκε να φύγουν, θα ήθελα να σας εκφράσω ε, τον περιόριστο σεβασμό μας και την ευγνωμοσύνη μας ε, για την τόσο αξιόλογη και αξιέπαινη δουλειά σας στη Μεσόγειο. Και τι παράξενο και ηρωνικό, η Νορβηγία δεν είναι καν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά παίρνει τόσο στα σοβαρά τις ανθρωπιστικές ανάγκες που υπάρχουν, που μερικές ε, φορές σκεφτόμαστε τι κρίμα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεχίστε παρακαλώ την καλή δουλειά. Γιατί τελικά το παράδειγμα μας θα επικρατήσει, το παράδειγμα σας θα επικρατήσει και θα εμπνεύσει πολλούς. Thank you, Cecilia. That was a long... Πριν από πάρα πολλά χρόνια είχαμε τους Vikings. Τέλος πάντων. Κύριε Γουίμπερν. Tack så mycket och tack så mycket herr Henriksen. Det var intressant att få se. Ε, Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ τον κύριο, ιδιαίτερα τον κύριο Χένριξεν, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα όσα είπε. Ε, τα πληρώματα έχω στο μυαλό μου, ε, στα οποία αναφερθήκατε κι εσείς. Ε, πρέπει να δούμε πιο προσεκτικά την κατάσταση, να δούμε πώς αυτά τα άτομα μπορούν να αντιμετωπίσουν τέτοια τραυματικά γεγονότα, οικογένειες νεκρές που επιπλέουν κλπ. Ε, η ψυχολογική πτυχή είναι πάρα πολύ σημαντική. Τα τελευταία δύο χρόνια έγιναν πολλά και αυτό που παρατηρούμε πλέον είναι ότι ε, υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις έρευνα και διάσωσης, αλλά θέλω να ρωτήσω τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει Πώς μπορούμε να αποφύγουμε να βαραίνει πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις στον εμπορικό στόλο. Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ε, υπευθυνότητα. Οι πιέσεις είναι πολύ σημαντικές, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς ε, μήνες. Ε, μιλήσατε και για τον ε, μιλήσαμε και για τον Ορισμό Εθνών και την δυνατότητα ενδεχομένω να πάρουμε την άδειά του προκειμένου να καταστρέψουμε τα σκάφη των διακινητών. Ε, κάτι τέτοιο στο παρελθόν ήταν ε, πολύ επιτυχές. οπότε ποια είναι η γνώμη σα γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους διερμηνείς και να μας, θα ήθελα να μας δώσουν λίγα λεπτά παραπάνω, αν γίνεται. Ευχαριστώ πολύ για την κατανόησή τους. Η Κορνίλια Ernst. Θα είμαι πολύ σύντομη. Εξ ονόματος της ομάδας της Αριστεράς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Παρακαλώ να το μεταβιβάσετε σε όλους τους συναδέλφους σας που δρούν τόπου. Πρέπει να πούμε ότι στην πράξη κάνουν πολύ περισσότερα από ό,τι κάνουν στο Συμβούλιο με τις άγονες συζητήσεις τους και τα μικρά αποτελέσματα. Υπάρχουν κάποια αντισταθμίσματα γιατί εσείς είσαστε εμπορικά πλοία. Έχετε τη δουλειά σας, δηλαδή η δουλειά σας δεν είναι η διάσωση ζώων σε τέτοια έκταση. Δηλαδή υπάρχει κάποια ε, οικονομική αμοιβή ε, και θέλω να προσθέσω στις ε, προτάσεις σας και συστάσεις σας κάτι ακόμα. Δηλαδή θα πρέπει να βρεθούν νομότυπες οδοί πρόσβαση στην Ευρώπη από αυτούς τους ανθρώπους ε, για να μην ακολουθούν αυτές τις φρικτές οδούς να μπορούν νόμιμα να ε, δικαιούνται είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος ε, Τζιρέκ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε κύριοι για την παρουσίαση και τις πληροφορίες που μας δώσατε. Ε, άκουσα με ενδιαφέρον τις ε, περιπτώσεις ε, επιθετικότητας που αντιμετωπίζετε στη θάλασσα από πλευράς ενόπλων, γιατί σπάνια ακούμε τέτοιες λεπτομέρειες επιθετικών κινήσεων, δηλαδή επιθέσεων εναντίον σας. Ίσως ε, θα, ε, θα μπορούσατε να μας δώσετε και άλλες τέτοιες ε, περιπτώσεις. Ευχαριστώ που είσαστε και πολύ σύντομος. Η Άννα Γκόμες. Ευχαριστώ που μας δίνετε όλα αυτά τα στοιχεία. Μας πείθετε ότι πολύ περισσότερα πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να κινητοποιήσει όλα τα μέσα της για να σώσει ζωές, γιατί είναι υποχρέωσή της κάτι τέτοιο. Εσείς τι άποψη έχετε που η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει μια αποστολή ΚΠΑ στη θάλασσα κατά της πειρατείας για την κοινή πολιτική ασφαλείας και άμυνας. Αλλά δεν είχε αποστολή ΚΠΑ για να σώσει ζωές. Δεν το θεωρεί πρώτη προτεραιότητα. Ούτε κατά των ε, διακινητών κάνει μια τέτοια αποστολή. Είναι, έχασε μια ευκαιρία, τραγική απώλεια, να χρησιμοποιήσει το ναυτικό των χωρών της ευρωπαϊκή Ένωσης στην υπηρεσία η εξυπηρέτηση αυτού του στόχου, που είναι η διάσωση ζώων. Στην απόφαση του Συμβουλίου, μάλιστα, αυτή η αποστολή θα πρέπει να έχει αυτό το καθήκον, να σώσει ζωές, γιατί αυτό είναι το δίκαιο της θάλασσας. Και αυτή η αποστολή πρέπει να εξυπηρετήσει αυτό το στόχο. Αλλά δεν είναι μια ευκαιρία που χάθηκε και δεν είναι γελίο αυτό που φαίνεται ότι υπάρχουν, υπάρχει το στρατιωτικό, το πολεμικό ναυτικό, ε, που όμως δεν εξυπηρετεί αυτό το υψηλό καθήκον της διάσωσης ανθρώπινων ζώων. Εγώ μίλησα σε κάποιον από τη Frontex και τους ρώτησα για το Μάρε Nostrum. Ποια είναι η νομική κατάσταση των εφοπλιστών. Εσείς ακούτε ας πούμε τα σήματα στον ασύρματο ε, για περιπτώσεις όπου ένα σκάφος κινδυνεύει. Αλλά μερικές φορές ε, τα σήματα αυτά, αυτά τα, τα μηχανήματα κλείνουν. Μπορείτε να μας περιγράψετε την πίεση που υφίστανται οι ναυτικοί σας. Μπορείτε να μιλήσετε έτσι, ξέρω εγώ, με, νούμερα λιγάκι. Για να καταλάβουμε την πίεση που τα μέλη σας υφίστανται. Ε, και να σκεγγραφίσουμε έτσι πιο ολοκληρωμένα την εικόνα. Η κυρία Μέρ είναι η επόμενη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τους προσκεκλημένους ομιλητές μας. Έχω κάποια πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Πρώτον, είναι προετοιμασμένα τα πληρώματα για τέτοιου είδους επιχειρήσεις έρευνα και διάσωσης. Ε, τι συμβουλές τους δίδεται. Ε, και κάποιος άλλος το ανέφερε, αλλά θα ήθελα περισσότερες λεπτομέρειες. Δεύτερον, σε ποιο βαθμό μπορούν οι εφοπλιστές να προστατεύουν τα πληρώματά τους από κίνδυνου στην θάλασσα, συμπεριλαμβανομένης και της τρομοκρατίας. Τρίτον, το κόστος ε, παρέμβασης, ε, η εκτροπής από την πορεία τους αυτών των σκαφών. finally, ε, ε, Σράια. Θα μιλήσω στα σουηδικά. Ε, θέλησα να παρέμβω και στην προηγούμενη μας ε, συζήτηση, ε, αλλά δεν τα κατάφερα. Ε, καταρχήν να δώσω όμως ε, τις ευχαριστίες μου στους δύο προσκεκλημένους μας. Κάνετε κάτι το οποίο θα έπρεπε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό λόγω αξίζεται το συγχαρητήριο μας. Επιπλέον υπάρχει και ένα κύμα άκρας δεξιάς, λαϊκιστικής άκρας δεξιάς στην Ευρώπη ε, που αρνείται την επιδείξη αλληλεγγύης μεταξύ όλων. Ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε ευρωσκεπτικιστές. Και όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να πω στην κυρία Βίμπερ τα εξή. Κριστίνα, τώρα που είδες όλα αυτά τα άτομα στο βίντεο, πιστεύετε ότι, πιστεύεις ότι ακόμα ότι είναι ε, δολοφόνη. Μου φαίνεται πραγματικά εκπληκτικό αυτό που είπε προηγουμένως. Μετά, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου αναφέρεται ότι η Frontex πρέπει να βοηθάει τα κράτη-μέλη να διαχειριστούν τις μεταναστευτικέ ροέ. Η Frontex θα πρέπει να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο. Η ερώτηση λοιπόν είναι τι θα γίνει με τον προπολογισμό ε, για τις επιχειρήσει, διάσωσης, ε, έρευνας και διάσωση στη Μεσόγειο. Ε, είναι επίσης ανησυχητικό το να καταρτίζουμε ένα κατάλογο ασφαλών χωρών. Δηλαδή θα πρέπει να ξεκινούμε από την υπόθεση ότι κάποιες χώρες είναι ασφαλείς και κάποιες όχι. Ε, δεν θα πρέπει να γίνεται εξέταση κατά περίπτωση για κάθε άτομο χωριστά. Έχω και άλλες ερωτήσεις αλλά δεν θέλω να πάρω άλλο χρόνο. Παρακαλώ να σκεφτόμαστε πάντα και πρώτα τους ανθρώπους. Ευχαριστώ. Κύριος Φερχόβεν και κύριος Χένριξεν, δεν χρειάζεται να απαντήσετε σε κάθε ερώτηση γιατί δεν έχουμε και τόσο χρόνο τόσο ή άλλως, προσπαθείτε να απαντήσετε τα βασικά στοιχεία, ε, το μήνυμα που σας έστειλαν οι ευρωβουλευτές. Ευχαριστώ. Θα απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις και ο Πάτρικ θα με συμπληρώσει. Για την ε, κατάρτιση των πληρωμάτων. Οι ναυτιλιακές εταιρείε είναι έτοιμες να το κάνουν αυτό και να εξοπλίσουν επίσης και τα πλοία. Τους προετοιμάζουμε έχουμε κατευθυντήρες γραμμές. Πρέπει να προετοιμάσουμε χώρους εισόδου. Ε, έχουμε πρακτικές κατευθυντήρες γραμμές δηλαδή. Δηλαδή όλο το πλήρωμα βάζουν ε, και προστατευτικά ε, και βάζουν και τις στόλες τους για να δείχνουν ποιος είναι ποιος και οργανώνουν τους ανθρώπους έτσι, με ομαδικό πνεύμα, γιατί ξαφνικά το εμπορικό πλοίο γίνεται ένα πλωτό, ας πούμε, ε, στρατόπεδο προσφύγων. Ε, έχουμε παιδιά, έχουμε γυναίκες της ίδιας οικογένειας, ας πούμε, άντρες κτλ. Υπάρχουν θέματα, ας πούμε, ε, υγιεινής, έχουμε κατευθύνσει αμέσως γι' αυτό, έχουμε μια υπηρεσία, ας πούμε, που απαντάει σε όλα τα επίγοντα, συνέχεια, να πάσα στιγμή. Έχουμε ε, επαφή, φέρνουν σε επαφή αυτά τα μέλη ε, με ψυχιάτρους, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν ε, τα ψυχολογικά προβλήματα που μπορεί να έχουν. Γιατί μπορεί να είναι πάρα πολύ έντονη αυτή η εμπειρία. Ειδικά όταν ψάχνεις τη θάλασσα, ας και βλέπεις παιδιά, ας πούμε, πτώματα παιδιών να πλέουν στη θάλασσα. Αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο να το ξεπεράσει κανείς. Λοιπόν, τι θα ήταν αρκετό. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεντρώνει α, τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή τη, του πόρου που έχει στη διάθεσή τη. Αυτό είναι ε, ευπρόσδεκτο. Επίση, μην ξεχνάμε ότι όλο και αυξάνεται ο αριθμό των, των, ανθρώπων ε, και περιμένουμε μεγάλη αύξηση του αριθμού των μεταναστών τους επόμενους μήνες. Γιατί τώρα ε, περάσαμε το ήσυχο ας πούμε, τμήμα της χρονιάς και τώρα ε, μπαίνουμε στην, στο high season ας πούμε. Και με βάση τις εκτιμήσεις της ΥΠΑ της, ε, θα έχουμε αύξηση 80% πάνω από 80%. Ε, για το αν θα ζητήσουμε αποζημίωση για τις επιχειρήσεις διάσωσης. Όχι, όχι, δεν θέλουμε ε, λεφτά, δεν θέλουμε αποζημίωση για κάτι τέτοιο. Θεωρούμε ότι είναι ηθικό μας και ανθρωπιστικό μας και νομικό μας καθήκον. Επίσης δεν θέλουμε αυτό να θεωρηθεί ως μόνιμη κατάσταση και να θεωρείτε ότι εμείς αποτελούμε τμήμα, ας πούμε, των πόρων που έχετε για να κάνετε αυτές τις ε, επιχειρήσεις ε, έρευνας και διάσωσης. Όχι, εμείς θα πληρώνουμε από τις τσέπες μας. Επίσης, δεχτήκαμε επιθέσεις. Ναι, σε ορισμένες περιπτώσεις απείλησαν ε, το μέλη του πληρώματό μας υπό την απειλή όπλου για να επιστρέψουν ας πούμε, το, τα σκάφη αυτά ε, στους διακινητές για να μπορούν να τα ξαναχρησιμοποιήσουν. Οι διακινητές το απείλησαν λοιπόν, ο συνάδελφος. Πολύ σύντομα, η συνεισηγήτρια είπε πώς θα βελτιωθεί ο συντονισμός ε, και με τον τρίτον αποσυδόν ε, Frontex. Είναι σημαντικό οι διαδικασίες αποβίβασης να γίνονται αποτελεσματικά είτε στην ξηρά ή σε άλλα σκάφη πολύ βασικό από επιχειρησιακής άποψης και όταν θέλουμε να συνεργαστούμε με τον τρίτονα. Επίσης, η αυτοπροστασία και η σύγκριση με την πειρατεία ε, είναι δύο διαφορετικά πράγματα εδώ. Ε, στην ε, Σομαλία είχαμε δεχτεί επιβίβαση ενόπλων. Εδώ όμως μπορεί να επιδεινωθεί το πρόβλημα γιατί είναι οργανωμένο έγκλημα. Ε, άνθρωποι δηλαδή που δεν θα φοβηθούν να πυροβολήσουν. Οπότε έτσι θα διακινδυνεύσουν περισσότερες ζωές και δεν θα βοηθήσουμε. Για την ε, ανταμοιβή μας, συμφωνώ με τον Στούρλα, Έχουμε στοιχεία σχετικά, αλλά δεν θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι εκεί αποσκοπούμε τα στοιχεία διαφέρουν, γιατί μπορεί να αλλάξει τη ρότα του το πλοίο για πολύ λίγο ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ε, είναι δύσκολο δηλαδή να δώσουμε νούμερα εδώ. Τώρα το λεπτό θέμα που θέσατε εσείς ε, σε σχέση με την αλλαγή σημάτων ε, DIS ε, δεν το ξέρουμε αν συμβαίνει αυτό το πράγμα οπωσδήποτε πρόκειται περί παρανομίας που πρέπει και να αναφέρεται αλλά μην ξεχνάμε ότι για πολλά σκάφη στην περιοχή είναι πολύ δύσκολο να το αποφύγουν γιατί πολλά σκάφη δραστηριοποιούνται δηλαδή ε, έχουμε ας πούμε από το Σουέζ ένα πέρασμα στη Μεσόγειο αλλά εκεί έχουμε πάρα πολλά σκάφη επίσης σκάφη που είναι στην ανοιχτή θάλασσα και δραστηριοποιούνται εκεί οπότε είναι δύσκολο να αποφύγουμε τέτοια περιστατικά αλλά αν γίνονται σκόπιμα θα πρέπει να ασχοληθούν και οι επαγγελματικές ενώσεις και τα μέλη μας ε, αυτά είναι κάποιες πρόσθετες ε, παρατηρήσεις που ήθελα να κάνω. Ευχαριστώ πολύ. Ε, νομίζω ότι εδώ τα μέλη μας εκτιμούν πάρα πολύ τον επαγγελματισμό με τον οποίο απαντήσατε σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ και εκ μέρους των εισηγητών είναι πολύ σημαντική αυτή η συνεισφορά και την εκτιμούμε όπως της αξίζει. Ευχαριστώ που αφιερώσατε χρόνο. Συνάδελφοι, ευχαριστώ ιδιαίτερα όλους όσους έμειναν μέχρι το τέλος. Πολύ το εκτιμούμε. Φτάζουμε στο τέλος λοιπόν αυτής της ε, συνεδρίασης. Δεν υπάρχουν διάφορα. Η επόμενη συνεδρίαση είναι 15 και 16 Ιουλίου. Ευχαριστώ πολύ.